θέσαμε να συνεχίσουμε την ε, αναγκαστική διακοπή στι 12.30, όπω προβλέπει δηλαδή το πρόγραμμα τη συνεδρίαση ακριβώ. Πρέπει να έχουμε ολοκληρώσει, λέει η Πρόεδρο, ε, στι 12.30 ακριβώ. Ελπίζουμε να βρεθεί μια λύση που κυρίω ε, να ικανοποιεί και τι δύο πλευρέ, αλλά και κυρίω και του διερμηνεί ω εργαζόμενου. Ξέρουμε ότι η εργασία σας είναι απόλυτα απαραίτητη και γι' αυτό ελπίζουμε πάρα αυτά να επιληθεί αυτή η διαμάχη, το οποίο ελπίζουμε και εμείς. Ε, ψηφίζουμε, λέει η Πρόεδρος, και τώρα ψηφίζουμε μια έκθεση πρωτοβουλίας και δύο ε, γνωμοδοτήσεις. Να προτείνω να ξεκινήσουμε καταρχάς με τις, ε, με τις ψηφοφορίες. Επτά Έκθεση πρωτοβουλίας για την, ε, τις γλώσσες στην ψηφιακή εποχή και έχουμε την κυρία Evans, η οποία ήταν η συγγήτρια εδώ. Θέλετε να πάρετε το λόγο, κυρία Evans. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και να ευχαριστήσω τους κοιόδες εισηγητής, του βοηθού μου και του συμβούλου τη ομάδα ε, και την Λίτ και αν ε, από την γραμματεία όλους ιδιαίτερο. Ε. με ο Νέδης Πλής, Ντάβιτ Χέξε και άλλοι. Ήταν τεράστιο ο όγκο τη δουλειά ο οποίο χρειάστηκε για την έκθεση πρωτοβουλία αυτή και θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ καλή σε ποιότητα και άλλωστε ε, πολύ, ή πιο πολλοί συμφωνούμε από αυτόν και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό και το γεγονό ότι εκδηλώθηκε τέτοιο ενδιαφέρον για το θέμα αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ Λεκή Πρόεδρο και περνάμε λοιπόν πάρα αυτά στι ψηφοφορίε. βασμό 14 ε, υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Τροπολογία 50. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Δεν φαίνεται τι ψηφίζετε εάν δεν σηκώνετε τα χέρια σας. Σας παρακαλώ να ξαναψηφίσουμε. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Η 51 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 54 υπέρ. Κατά. Αποχές έγκρινεται. 53 υπέρ. Κατά. Αποχές έγκρινεται. Συμβαστική 9 υπέρ. Κατά. Αποχές έγκρινεται. 61 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 10 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ήτρε 50 υπέρ. 15 υπέρ κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ήτρε 16 υπέρ. Κατά. Έλεγχος ζητείτε. Πολύ ωραία. Λέει ο πρόεδρο να ελέγξουμε τη 15. Ψηφίζουμε παρακαλώ ηλεκτρονικά. Είναι Πέρασα. 15 υπέρ, 8 κατά. Εγκρίνεται. Ήτρε 16 υπέρ, κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ήτρε 17 υπέρ, κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 11. Συμβαστική 11 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 69 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 70 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 12 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ας ελέγξουμε λοιπόν και τη συμβαστική 12 αφού το επιθυμείτε. Πέρασε. 13 υπέρ, 10 κατά εγκρίνεται. Και περνάμε τώρα στην 77 υπέρ. Κατά. Αποχές. Έγκρινεται. 78 υπέρ. Κατά. Αποχές. Έγκρινεται. 79 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 13 υπέρ. Κατά. Αποχές. Έγκρινεται. 83 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 86. Α, συγγνώμη, 87. Ζητάει, συγγνώμη, πρόεδρος, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 88 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 89 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 15. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 91. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 92. Υπέρ. Κατά. Άποχες εγκρίνεται. Συμβαστική 16 υπέρ. Κατά. Άποχες εγκρίνεται. Ήτρε 19 υπέρ. Κατά. Αποχές έγκρινεται. Ήτρε 20 υπέρ. Κατά. Αποχές έγκρινεται. Ήτρε 6 υπέρ. Κατά. Άποχες έγκρινεται. 97 υπέρ. Κατά. Άποχες απορρίπτεται. Συμβαστική 17 υπέρ. Κατά. Άποχες έγκρινεται. 102 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται 101. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 104. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ήτρε 7. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Ήτρε 10. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Συμβαστική 18. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. 81 υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Έλεγχος. Για την 81. Πέρας. 13 υπέρ, 11 κατά. Εγκρίνεται. 64 υπέρ. Κατά. Απόχες. Έλεγχος παρακαλώ για την 64. Ψηφίζουμε. Πέρας. 15 υπέρ, 9 κατά, εγκρίνεται. 111 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 112 υπέρ, κατά, αποχές, ε, απορρίπτεται. Έλεγχος. 112 παρακαλώ. Πέρας. 12 ψηφία, 12 υπέρ, 12 κατά, απορρίπτεται άρα. 113 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 116 υπέρ, κατά, αποχές, Εγκρίνεται. 118 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 119 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 120 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 121 υπέρ. Κατά. Άποχες. Έλεγχος παρακαλώ για την 121. υπέρα. 13 υπέρ, 12 κατά. Εγκρίνεται. 122 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 123 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 125 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 19 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 314 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 20 υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Συμβαστική 21 υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Η 4 υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Συμβαστική 1 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 9 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 11 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 3 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 18 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 4 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ήτρε έψιλον, ε, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 5 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 6 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ήτρε εμ μη υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 7 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική. Α, συγγνώμη, τροπολογία 33. Λέει πρόεδρο υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 34 υπέρ. Κατά. Αποχές ε, ε, εγκρίνεται. 35 υπέρ. 34 θέλετε έλεγχο για 34 παρακαλώ να γίνει. Πολύ ωραία ηλεκτρονική ψηφοφορία για την 34. Πέρας. ψηφία. Απορρίπτεται. 35. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 36. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 8 υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρινέται. 41 υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. 42 υπέρ. Κατά. άποχε, Απορρίπτεται. 43 και ήτρε εν. Νι. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. 44 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 45 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 46 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Προφορική τραπολογία. 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ήτρε 1. γιώτα Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ήτρε Κάπα. Υπέρ. Κατά.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 κατά αποχές εγκρίνεται. Τροφολογία 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και περνάμε τώρα στην τελική ψηφοφορία με ονομαστική κλίση και έναρξη της ψηφοφορίας παρακαλώ. Πέρασε. 22 ψήφοι υπέρ, καμία ψήφος κατά Τέσσερις αποχές, ομόφωνα λοιπόν εγκρίνεται. Και συγχαρητήρια στην εισηγητρία. Θα περάσουμε τώρα στο σημείο 8 της σημερινής της διάταξης, στην ε, γνωμοδότηση για την ε, όθηση της ανάπτυξης και της συνοχής σε παραμεθόριες περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, εισηγητής μας ήταν ο κύριος Σεγοράκης. Δεν είναι παρόν. Δεν θα του δώσω λοιπόν το λόγο. Μπορούμε πάρα αυτά να περάσουμε στην φορεία και να ξεκινήσουμε με την τροπολογία 1 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρινέται. Τροπολογία 2 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρινέται. 3 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρινέται. 4 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 1 υπέρ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 Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 25 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 27 υπέρ. 26 συγγνώμη υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 27 υπέρ. Κατά. Αποχές ε, απορρίπτεται. Συμβαστική 3 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Και περνάμε στην τροπολογία 35 υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 4 υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. 36 υπέρ. Κατά. Άποχες. Απορρίπτεται. 38 υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. 39 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 40 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 41 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 5 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 51 υπέρ. Κατά. Αποχές Εγκρίνεται. 52 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 53 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 54 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 55 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 56 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 6 υπέρ Κατά. Αποχές. Έγκρινεται. Τροπολογία 62. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Έγκρινεται. 63. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Έγκρινεται. 64. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Έγκρινεται. 65. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Έγκρινεται. 66. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Έγκρινεται 67. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Έγκρινεται 68. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Έγκρινεται 69. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Έγκρινεται 70. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Έγκρινεται 71. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Έγκρινεται και τώρα περνάμε στην τελική ψηφοφορία με ονομαστική κλίση και έναρξη της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας λοιπόν. Πέρασε. 24 ψήφοι υπέρ, 0 κατά, μία αποχή, ομόφωνη η έγκριση, συγχαρητήρια στον εισηγητή. Περνάμε τώρα στο σημείο 9 της ημερήσιας διάταξης για την γνωμοδότηση για την τη θάσευση της παγκοσμιοποίησης εμπορικές πτυχές. Ο συνάδελφος της Άμετ Ντίμεκ είχε το, ρόλο το του εισηγητή και έχει και το λόγο για να κάνει σχόλιο. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους για τη σύνταξη αυτής της νομοθετικής γνωμοδότησης. Βρήκαμε τη σωστή ισορροπία για να τονίσουμε την πολιτιστική διάσταση όταν μιλάμε για την ε, αξιοποίηση της ε, ε, παγκοσμιοποίησης. Όλες τις ε, πολιτιστικές πτυχές στα πλαίσια της ελευθερίας έκφρασης και πλουραλισμού. Καταφέραμε να βάλουμε αυτές τις αρχές όταν μιλάμε για την παγκοσμιοποίηση. Σας ευχαριστώ πολύ και τώρα περνάμε στην ψηφοφορία. Τροπολογία 41, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 42, υπέρ. Κάτα. Αποχές εγκρίνεται. 43 υπέρ. Συγγνώμη, λέει η πρόεδρος, η 44 και τη 43 δεν την ψηφίζουμε. 44 λοιπόν υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 45 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 3 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Και περνάμε στη 53 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 54 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε στην 58 υπέρ κατά αποχές. Ας το ελέγξουμε παρακαλώ. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά για την 58. Πέρασε. 13 ε, ψήφοι κατά, 12 υπέρ. Απορρίπτεται. Τροπολογία 60 λοιπόν. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 68 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 61 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 5 υπέρ. Κατά αποχές ε, εγκρίνεται. Πάμε στην 67 ε, υπέρ. Κατά. Αποχές. Μου φαίνεται ότι εγκρίνεται, αλλά στο ελέγξουμε κιόλα. Έναρξη ψηφοφορία. Πέρας. 15 υπέρ, 9 κατά εγκρίνεται. Συμβαστική 6 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται 74 υπέρ κατά αποχές έγκρινεται 75 υπέρ κατά αποχές έγκρινεται υπέρ 65, 75 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 76 υπέρ κατά αποχές έγκρινεται 77 υπέρ κατά αποχές έγκρινεται ε, ε συμβαστική 7 υπέρ κατά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 Έναρξη ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Πέρας. Τα 4 υπέρ, 9 κατά. Εγκρίνεται. Ζητώ συγγνώμη. 20 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 1 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 24. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 2 υπέρ. Κατά. Αποχές έγκρινεται. 29 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 30 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 31 υπέρ. Κατά. Άποχες εγκρίνεται. 32 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 33 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 34 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 35 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ας ελέγξουμε παρακαλώ 35. Ψηφίζουμε. 15 υπέρ, 10 κατά εγκρίνεται. Και περνάμε στην 36 υπέρ. Κατά. Αποχές. Έγκρινεται. 37 υπέρ. Κατά. Αποχές. Έγκρινεται. 38 υπέρ. Κατά. Αποχές. Έγκρινεται. 39 υπέρ. Κατά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 Και τώρα περνάμε στην τελική ψηφοφορία με ονομαστική κλίση και ψηφίζουμε λοιπόν τώρα. Πέρασε. 25 ψήφοι υπέρ, καμία ψήφος κατά, καμία αποχή, ομόφωνη έγκριση, συγχαρητήρια. Αυτά δεν τα βλέπουμε συχνά. Τέτοια αποτελέσματα δηλαδή. Έχουν καταφτάσει προσκεκλημένοι μας. Policy Department B und Kommission. Και του περάσουμε στο σημείο 10 της σημερινής διάταξης, ε, θα χρειαστεί να περιμένουμε λιγάκι μέχρι να διαπιστώσουμε αν έχουν καταφτάσει η προσκεκλημένοι μας. Και θα συνεχίσουμε παρά we start? So, Αγαπητοί συναδελφοί, να περάσουμε στο 10 τη ημερήσιας διάταξης. Ανταλλαγή απόψεων με την Επιτροπή και παρουσίαση μελέτης του θεματικού τμήματος για το πρόγραμμα Erasmus όπως ξέρετε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, παρουσίασε το νέο της πρόγραμμα για το μέλλον του πρόγραμματος Εράσμους. Ωστόσο, το πρόγραμμα Εράσμους μετά την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πλέον δεν φέρει το πρόσημο σύν Erasmus Plus. Σήμερα λοιπόν θα συζητήσουμε, θα συνεχίσουμε την ανταλλαγή απόψεων και θα έχουμε δύο τμήματα στην όλη συζήτηση. Καταρχάς θα παρουσιάσουμε την σχετική μελέτη του θεματικού τμήματος. Να καλωσορίσουμε την Άννα Γράφε που ε, εκπροσωπεί το ανεξάρτητο ερευνητικό ίδρυμα Παντέια και τον κύριο Μπούνχοφ, ο οποίος την ε, συνοδεύει και επίσης ε, είναι στη διάθεσή μας για τυχόν ερωτήματα για το νέο πρόγραμμα, τη νέα γενιά προγραμμάτων, έχει κάνει σχετικές μελέτες ε, για θέματα τα οποία μας απασχολούν ε, ιδιαίτερως και εμάς σε ό,τι αφορά και τις νέες ε, προτάσεις. Σε ό,τι αφορά, για παράδειγμα, την απλοποίηση, τον κοινοβουλευτικό έλεγχο και πολλά άλλα θέματα. Να σας συστήσω λοιπόν να διαβάσετε την μελέτη και στη συνέχεια θα περάσουμε στην παρουσίαση της νέας πρότασης από την Επιτροπή την ίδια. Να καλωσορίσω τον κυρία Έριξον του που είναι δευθύντρια για την εκπαίδευση για το Erasmus Plus από τους κόλπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά θα ξεκινήσουμε, όπως σας είπα, με την κυρία Άμπερ Φαντερ Χράφ, που θα έχει 10 λεπτά στη διάθεσή της για να μας παρουσιάσει τα αποτελέσματα της μελέτης. Ξέρω ότι δεν είναι μεγάλο το χρονικό διάστημα. Κάντε μια απόπειρα και σίγουρα και στις συζητήσεις, ερωτήσεις και τη συζήτηση που θα ακολουθήσει θα διευκρινίσουμε πολλά άλλα ζητήματα. Ευχαριστώ. Thank you. Good morning everyone. Καλημέρα. Λέγομαι Άμπερ Βαντεγκράφ από το Γραφείο Ερευνών της Παντέια στην ε, Ολλανδία και θα παρουσιάσω αυτή τη μελέτη για το Erasmus Plus ε, που το ζήτησε η Επιτροπή Πολιτισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα εστιάσουμε στα βασικά πορίσματα και σε βασικά συμπεράσματα σε αυτή την παρουσίαση. Ο στόχος της μελέτης ήταν τριπλός. Καταρχάς, ε, να εξετάσουμε τα αποτελέσματα του Erasmus Plus, ε, βασιστήκαμε σε ερευνητικά στοιχεία που είχαμε σε Ευρωπαϊκή Ένωση και σε εθνικό επίπεδο, καθώς και τις εμπειρίες από το νέο σχεδιασμό προγράμματος. Ε, επίσης, ε, τη διαδικασία λήψης των αποφάσεων στο Erasmus Plus και κατά πόσον χρειάζεται μια διαφορετική διαδικασία αποφάσεων για την εφαρμογή του προγράμματος. Ο τρίτος στόχος είναι να φτάσουμε σε συμπεράσματα για την επόμενη γενιά προγράμματος ε, θα κάνω ένα προβληματισμό επίσης για την ενδιάμεση αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε αυτή τη μελέτη. Κάναμε έρευνα με βάση τη βιβλιογραφία και κάποιε συνεντεύξει σε Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικό επίπεδο. Το βασικό αποτέλεσμα είναι ότι το Erasmus Plus ε, είναι καλό πρόγραμμα, έχει υψηλή προστιθέμενη αξία σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο και επιτρέπει διάφορα σχέδια και προγράμματα να εφαρμοστούν. Υπάρχει μεγάλη ζήτηση για το πρόγραμμα. Αυτό δείχνει και η μεγάλη απορρόφηση των κονδυλίων, σχεδόν 100% και υπάρχει το εξή φαινόμενο, ότι η υποβολή των αιτήσεων, οι αιτήσει μάλλον, ε, είναι όλο και πιο ποιοτικέ, αλλά τα ποσοστά επιτυχία ε, μειώνονται. Ε, Επομένω, αυτά είναι τα όρια του το πρόγραμμα Εράσμους. Η μελέτη αυτή εξετάζει και το βαθμό στον οποίο τα, οι στόχοι έχουν, από τον νέο σχεδιασμό έχουν υλοποιηθεί. Το νέο πρόγραμμα έχει τρεις ε, βασικές ε, δράσεις ε, σε διάφορους τομείς που συμπληρώνουν διάφορες δραστηριότητες. Τα βασικά θέματα είναι ορατότητα, μη αποκλεισμή, διατομιακή συνεργασία, απλούστευση του προγράμματος, αποτελεσματικότητα κτλ. Υπάρχει περιθώριο με βάση αυτές τις αρχές να υπάρξει μεγαλύτερη βελτίωση. Ξέρετε όλοι, φαντάζομαι, την ενδιάμεση αξιολόγηση Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ε, τεράστια μελέτη αυτή. Ε, με βάση τη μελέτη μας κάνουμε και ένα προβληματισμό για αυτή την ε, μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σε μεγάλο βαθμό συμφωνούμε με τα απορίσματα της διάμεσης αξιολόγησης τα ξέρετε κάποια από τα βασικά πορίσματα. Καταρχάς, ε, πώς θα φτάσουμε στις διάφορες ομάδες, είναι πρόβλημα. Ε, η κατανομή του προϋπολογισμού ε, γίνεται με βάση την παλιά κατανομή. Επίσης, η διαδικασία των αιτήσεων είναι μακρά, περίπλοκη, επαχθής. Ο μηχανισμός χρηματοδότησης φοιτητικών δανείων δυστυχώ δεν ήταν στο ύψος των προσδοκιών και υπάρχει και σε ό,τι αφορά την μάθηση των ενηλίκων, υπάρχει κατακαιρματισμός. Υπάρχουν διάφορα άλλα σημεία που, που καλύπτονται στην διάμεση αξιολόγηση, αλλά όχι στη δική μας μελέτη. Ε, μπορούμε να, με βάση τις μελέτες που κάναμε να δώσουμε κάποιες αποχρώσεις και μια νέα προοπτική. Ε, παρότι η ευθυγράμμιση ανάμεσα στα σχέδια και τις ευρωπαϊκές προτεραιότητες ε, δεν είναι απόλυτη. Παρ' όλα αυτά, οι προτεραιότητες είναι ευρείε και θέλουμε ε, οι, ε, οι δικαιούχοι να συμμετέχουν στα προγράμματα με βάση ανάγκες τους. Υπάρχει χαμηλό επίπεδο καινοτομία. Ε, αυτό αναφέρεται, αλλά αυτό δεν το βρίσκουν σωστό οι δικαιούχοι. Δεν συμφωνούν δηλαδή οι δικαιούχοι. Σε ό,τι αφορά τον αθλητισμό υπάρχουν πάρα πολλέ προτεραιότητες ε, και αμφισημίε. Ε, σωστό είναι αυτό το συμπέρασμα σε κάποιο βαθμό τη ενδιάμεση αξιολόγηση, Ε, αλλά αυτό δεν είναι κατά αναγκαία δυναμία. Ε, με αυτόν τον τρόπο διάφορα προγράμματα ε, που υποστηρίζουν διάφορους στόχους του Εράσμους ε, προωθούνται και υποστηρίζονται. Υπάρχουν άλλες πτυχέ που δεν τις έχουμε σκεφτεί πολύ. Παραδείγματο χάρη ε, το σύστημα έχει στενή εστίαση στι δραστηριότητε Ζαμονέ. Ε, συλλέγονται πάρα πολλά δεδομένα. Ε, εμείς πιστεύουμε ότι υπάρχουν και άλλες πτυχές ε, στις οποίες η τρέχουσα μελέτη ε, έχει φτάσει σε τελείως διαφορετικά πορίσματα. Το Erasmus Plus εφαρμόζεται χρησιμοποιώντας τα ετήσια προγράμματα εργασίας, τα οποία χρησιμοποιούνται, αναπτύσσονται χρησιμοποιώντας ε, τις, τη διαδικασία των εφαρμοστικών πράξεων και τη διαδικασία της εξέτασης. τα εξετάζει τα συντάσσει η ετήσια η Κομισιόν ε, και έχει διάφορους ε, τομείς εστίασης, ε, την κατανομή του προϋπολογισμού για διάφορες βασικές δράσεις, τομείς κτλ. Το πώς κατανέμονται τα κονδύλια στις εθνικές, στους εθνικούς οργανισμούς. Επομένως, όταν υπάρχει μεγαλύτερη ευθυγράμμιση με τις αιτήσεις αυτές προτεραιότητες, θα πάρουν αυτά τα εκεί θα πέσουν και τα περισσότερα κονδύλια. Γενικά η εφαρμογή θεωρείται ότι πηγαίνει καλά. Οι πάλι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, και οι εθνικοί δικαιούχοι είπαν ότι γενικά υπάρχει καλή σχέση εργασίας και υπάρχει ανταπόκριση στις εθνικές ανάγκες. Ένα σημείο συζήτησης στη διαδικασία λήψη των αποφάσεων τη Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η εφαρμογή των ε, κατεξοδότηση και εφαρμοστικών πράξεων. Πότε θα εφαρμόσουμε τι ΜΕ και πότε τι ΔΕ. Ε, αυτό το λέει ξεκάθαρα, το, τα λένε ξεκάθαρα τα κείμενα, αλλά στην πράξη είναι πιο δύσκολα τα πράγματα. Ξέρετε ότι με τι κατεξοδότηση πράξει εμπλέκονται οι νομοθέτε. Ενώ ε, στην άλλη περίπτωση ε, εμπλέκεται η Επιτροπή Προγράμματο. Ε, οι αιτήσει προτεραιότητε είναι ένα παράδειγμα τέτοιων προβλημάτων όπου η, αίτηση, όπου η εφαρμογή ε, της μίας ή της άλλης διαδικασίας δεν είναι τόσο απλή. Ε, οι αιτήσει προτεραιότητες πρέπει να εφαρμοστούν βεβαίως, έτσι μπορούμε να το δούμε από τη μία. Από την άλλη, ε, μπορούμε να θεωρήσουμε ότι είναι πιο πολιτικές ή πιο στρατηγικές αποφάσεις. Επομένως, το επιχείρημα υπάρχει ότι για αυτέ τι αιτήσει προτεραιότητε μπορούν και η κατεξιοδότηση και οι εφαρμοστικέ πράξει να εφαρμοστούν. Ε, Εναλλακτικέ ε, διαδικασίε αποφάσεων είναι δύσκολο να εφαρμοστούν. Υπάρχουν περιορισμοί λόγω της ε, διαθεσμικής συμφωνίας του 16 και της κοινή ε, συνεννόησης. Ε, σε πολλέ περιπτώσει, όμω, οι εφαρμοστικέ πράξει είναι ο κατάλληλο μηχανισμό για την εφαρμογή του Erasmus Plus. Ε, τον, το θέμα των ετήσιων προτεραιοτήτων και η θέση του στα ετήσια προγράμματα εργασία είναι ένα θέμα συζήτηση. Μπορούμε να κάνουμε δύο επιπλέον συστάσεις ό,τι αφορά την διαδικασία λήψη των αποφάσεων στο Erasmus Plus. Θα μπορούσαμε να ορίσουμε πιο σαφώς ε, ποιε πτυχέ του προγράμματος ε, εμπίπτουν Στι εκτελεστικές και ποιες εφαρμοστικές ε, και ποιες καταξιοδότηση πράξεις όταν συντάσσουμε τη βασική πράξη ε, για να μην έχουμε να χρησιμοποιούμε δύο διαδικασίες στο μέλλον. Επίσης, δεύτερον, να σκεφτούμε πολύ προσεκτικά το, τη θέση και το ρόλο των ετήσιων προγραμμάτων εντός των ετήσιων προγραμμάτων εργασίας και πώς θα αποφασίζουμε για αυτό το σημείο. Μετά από αυτά τα βασικά πορίσματα της μελέτης, θέλω να φτάσω στις ε, συστάσεις και τα συμπεράσματα στα οποία φτάσαμε. Το Erasmus Plus που σας είπα τα πάει καλά. Υπάρχει υψηλή προστιθέμενη αξία για όλους τους εμπλεκόμενους. Το νέο πρόγραμμα, ο νέος σχεδιασμός έχει βοηθήσει για την καλύτερη ορατότητα, απλουστευμένο προγραμματισμό, ε, διατομιακή συνεργασία, μη αποκλεισμού, αποτελεσματικότητα και καλύτερο προσανατολισμός στα προγράμματα. Παρ' όλα αυτά μπορούμε να κάνουμε βελτιώσεις. Ε, Υποστηρίζουμε τις, ε, την αξιολόγηση ευρωπαϊκής ε, μελέτης. Ε, φτάνουμε όμως και σε διάφορες συστάσεις. Ε, αναφέραμε κάποιες από αυτές εδώ. Ένα πρώτο βήμα θα ήταν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να κάνει κάτι, να σκεφτεί και να αποφασίσει τις βασικές προτεραιότητες για το Erasmus+. Είναι ευρύ πρόγραμμα ε, και φυσικά είναι πεπερασμένοι οι πόροι του και γι' αυτό θα πρέπει να γίνουν επιλογές. Με βάση την έρευνα που κάναμε, κάποιες βασικές συστάσεις του προγράμματος ε, προκύπτουν. Ε, θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη συμμετοχή και προσπελασιμότητα, μεγαλύτερη χρηματοδότηση στον τομέα της νεολαίας και καλύτερη στοχοθέτηση των μικρότερων οργανώσεων ε, και των νεοφερμένων, να μειώσουμε την περιπλοκότητα και το διοικητικό άχθος. Θα μπορούσαμε λοιπόν ε, να αντιμετωπίσουμε αυτά τα προβλήματα. Εάν θέλετε να δείτε περισσότερα συμπεράσματα και συστάσεις, ε, μπορείτε να διαβάσετε την εκθεσή μας. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Φανερχράφ για την παρουσίαση αυτής της μελέτης, η οποία ήδη νομίζω μας υποδεικνύει που θα πρέπει να επιδείξουμε προσοχή σε ό,τι αφορά το νέο πρόγραμμα και να ευχαριστήσουμε ιδιαιτέρως και για τις προτάσεις τις οποίες μας ε, κάνατε για το τι θα πρέπει να βελτιώσουμε στα νέα προγράμματα. Νομίζω ότι μας ε, διευκρινίσατε τι ισχύει για τις πράξεις κατά εξουσιοδότηση και τι μπορεί να κάνει το Κοινοβούλιο για να καταλήξουμε σε μια πιο άνετη κατάσταση, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τη λήψη πολιτικών αποφάσεων. Γιατί σε ό,τι αφορά τι εκτελεστικέ πράξει, διαπιστώνουμε ότι σε πολλέ περιπτώσει δεν είναι αμυγό τεχνικά τα θέματα, αλλά κάνουν και μια ιεράρχηση, μια, ε, ένα καθορισμό των προτεραιοτήτων και αυτό προφανώ είναι στον τομέα αρμοδιοτήτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σα ευχαριστώ και νομίζω ότι για να α, μεγιστοποιήσουμε, αν θέλετε, την αποτελεσματικότητά μα, θα δώσουμε το λόγο παραστά στην κυρία Έριξον να μα παρουσιάσει την καινούργια πρόταση για να τα συζητήσουμε όλα αυτά από κοινού στη συνέχεια. Όλοι λοιπόν θα έχετε δει το πρόγραμμα αυτό. Διαπιστώσαμε μεν ότι υπάρχει αύξηση των ε, κονδυλίων. Αυτό είναι φυσικά ευχάριστο. Αλλά όχι αυτή που είχαμε ζητήσει ως Κοινοβούλιο. Έχουμε και το ψήφισμα για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Είχαμε ζητήσει τριπλασιασμό των πόρων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει διπλασιασμό των κονδυλίων και αν συνυπολογίσουμε και τον πληθωρισμό δεν είναι φυσικά διπλασιασμένο το ποσό, αλλά 26 δις, το οποίο ουσιαστικά θα ήταν ε, αυτό που θα αναλογούσε στο πρόγραμμα και στη συνέχεια αυτού. Δεν μπορούμε λοιπόν να θεωρήσουμε ότι είμαστε ικανοποιημένοι. Και κοιτώντα περαιτέρω και την πρόταση για το πρόγραμμα Εράσμους, διαπιστώνουμε ότι ενώ έχουν διευρυνθεί κατά πολύ μάλιστα η στόχη, η στοχοθεσία σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα Εράσμος. Το ίδιο το πρόγραμμα Εράσμος έχει καταστεί πολύ πιο ασαφές. Πολύ πιο ασαφές σε σχέση με την προηγούμενη πρόταση. Και θα πρέπει το Κοινοβουλίο λοιπόν να εξετάσει το κατά πόσο να... Το Κοινοβούλιο ουσιαστικά δίνει λευκή επιταγή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει λοιπόν να τα συζητήσουμε αυτά σοβαρά. Κατά πόσον ε, οι συγκεκριμένε προτάσεις όπως ήταν στο παλιό πρόγραμμα ήταν πολύ καλύτερες ε, για την ιεράρχηση των προτεραιοτήτων μας. Παρά την γενική αυτή, την γενικόλογη πρόταση, τουλάχιστον αυτή την εντύπωση έχουμε εκ πρώτης όψεως. Ε. Γι' αυτό λοιπόν Αυτές είναι οι δικέ μου πρώτες παρατηρήσεις. Ε, στη συνέχεια θα μας πείτε και εσείς τι πιστεύετε. Κυρία Έρεξον, παρά το λόγο 10 λεπτά και πείτε μας τι αλλάξατε και γιατί. Σίγουρα πρόκειται για μια μεταξέλιξη, όχι πραγματικά για μια επαναστατική διαμόρφωση του προγράμματος. Αλλά πείτε μας λοιπόν τι σας όθησε να κάνετε τις προτάσεις που κάνετε από πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στη συνέχεια προσβλέπω και σε μια εκτενή συζήτηση για την οποία έχουμε προβλέψει πολύ χρόνο. Κυρία Έριξον. Thank uh, Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, από τα μέλη του Κοινοβουλίου. Ε, διότι χαρά για μένα που θα μπορέσω να σας παρουσιάσω την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το νέο πρόγραμμα Erasmus, η οποία εγκρίθηκε τον προηγούμενο Μάιο. Ε, γνωρίζετε ποιο είναι το πολιτικό πλαίσιο και είναι εξαιρετικό που έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε ένα πρόγραμμα το οποίο, έχει, το οποίο η αξία έχει αναγνωριστεί ε, για την νεολαία, για την εκπαίδευση και ακριβώς επειδή έχει αναγνωριστεί η αξία του, ε, του έχει δοθεί και μια μεγάλη όθηση. Θα ήθελα να ευχαριστήσω, αν και καθυστερημένα, ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την υποστήριξη και για τη δυνατότητα ότι μας βοηθήσατε να γιορτάσουμε τα 30 χρόνια του Εράσμους πέρυσι. σε αυτήν την ε, εκδήλωση στις 30 Ιουνίου ε, στο Στρασβούργο πέρυσι. Ήταν μια εκδήλωση η οποία έδωσε δημοσιότητα και έδωσε τη δυνατότητα ε, αργότερα να προετοιμάσουμε και εμείς και να παρουσιάσουμε αυτήν την φιλόδοξη πρόταση για τον νέο Εράσμος. Γνωρίζετε ότι η δημοσιοποίηση της πρότασής μας έγινε ακριβώς την ίδια στιγμή με την έναρξη συζητήσεων πολύ σημαντικών για τον τομεί πολιτικής, της εκπαίδευσης, της έρευνας. Επομένως, τις διάφορε επιδιώξεις, τις διάφορες φιλοδοξίε προσπαθήσαμε να τις μεταφέρουμε και στην πρόταση του προγράμματος. Έχει αναγνωριστεί ως εμβληματικό το πρόγραμμα Εράσμού. και νομίζω θα ήταν σκόπιμο να ακούσουμε ορισμένα αριθμητικά στοιχεία. Έχουν γίνει πολλέ αξιολογήσει τύπου για του δικαιούχου και εκείνου που αξιοποίησαν το Εράσμο. Θα αναφέρω μόνο δύο στοιχεία που μιλούν από μόνα του, κατά την άποψή μου. Το ένα στοιχείο είναι ότι εκείνοι που έχουν συμμετάσχει στο Εράσμος έχουν ε, καλύτερη πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Έχουμε διαπιστώσει ότι διπλασιάζεται η δυνατότητά τους να βρουν δουλειά ένα χρόνο μετά την αποφύτισή τους. Και όχι μόνο αυτό, και στην ε, μη τυπική εκπαίδευση το βρίσκουμε αυτό. στην μη τυπική εκπαίδευση είναι 35% περισσότερε οι πιθανότητε σε σχέση με κάποιον ο οποίο δεν είχε παρακολουθήσει πρόγραμμα Εράσμου. Υπάρχει επίση και ένα άλλο πλεονέκτημα του Εράσμου, ότι ενώνει την Ευρώπη, ότι ερχόμαστε μαζί και ε, ε, το διαπιστώνουμε αυτό στις φιγρομετρήσεις εκείνων που συμμετείχαν σε μια ανταλλαγή Εράσμους, αισθάνονται περισσότερο Ευρωπαίοι και δηλώνουν ότι ε, έχει αυξηθεί επίσης και η ανοχή τους προς τη διαφορετικότητα, η κατανόησή τους προς τη διαφορετικότητα. Γνωρίζουμε επίση ότι το πρόγραμμα Erasmus έχει θετικέ επιδράσει και στα διάφορα ευρήματα που, γίνονται, που ανοίγουν προ τα έξω και προ τη διεθνή πραγματικότητα. Η αξιολόγηση του Erasmus έχει κρατήσει πάνω από ένα χρόνο και προσπαθήσαμε σε αυτή την περίοδο προετοιμασίας να συμμετάσχουν όλοι όσοι έχουν οποιαδήποτε σχέση και ενδιαφέρον για το πρόγραμμα του Εράσμου. Αυτό προφανώ περιλαμβάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά επίση και τι εθνικέ αρχέ, τα διάφορα ιδρύματα κτλ. Αξιοποιήσαμε εκθέσεις πολλές από την ε, επιτροπή σας. Είχαμε ένα εκατομμύριο απαντήσεις στη δημόσια διαβούλευση, είναι εντυπωσιακός ο αριθμός. Και τα συμπεράσματα αυτή τη διαβούλευση ταιριάζουν πολύ και με τα συμπεράσματα και με τα ευρήματα της έρευνας που μόλις μας παρουσιάστηκε, γι' αυτό και δεν θα επανέλθω. Όμως, όπως είπατε κι εσείς, υπήρξε μεγάλη ε, υποστήριξη στο να υπάρξει συνέχεια, ακριβώς επειδή το πρόγραμμα ήταν επιτυχημένο. Η συζήτηση που είχε γίνει την προηγούμενη φορά ε, ήταν δύσκολη γιατί έπρεπε να συνενώσουμε 7 διαφορετικά προγράμματα. Όμω τώρα πια έχει κυλήσει και το νερό στα βλάκια και διαπιστώνουμε ότι ε, οι συμμετέχοντες και αυτοί με τους οποίους συζητούμε επιθυμούν να συνεχίσουν τα πράγματα με τρόπο πολύ παρόμοιο. Γι' αυτό και εμείς η πρότασή μας είναι μια μετεξέλιξη όχι μια επαναστατική αλλαγή. Προτείνουμε να κρατήσουμε την ίδια αρχιτεκτονική και στο μέλλον, προτείνουμε να παραμείνει ίδιο το πεδίο εφαρμογή του προγράμματος και ε, το, οι διαδικασίες για την ε, εφαρμογή του να παραμείνουν πάνω κάτω οι ίδιες. Με λίγα λόγια δηλαδή, να κρατήσουμε αυτό το μοντέλο με τις εθνικές αρχές υλοποίησης που έχει αποδείξει την αποτελεσματικότητά του. Σε αφορά τη δομή, την αρχιτεκτονική, ε, διαπιστώνουμε ότι υπάρχει υποστήριξη για το να κρατήσουμε τους τρεις πυλώνες. Είναι ξεκάθαροι, έχουν απλούς, είναι εύκολο να τους αντιληφθεί κανείς. Δηλαδή, την κινητικότητα, την συνεργασία μεταξύ ιδρυμάτων σε οποιοδήποτε τομέα και τρίτος πυλώνας, μικρότερος, η ανάπτυξη, η υποστήριξη στην ανάπτυξη πολιτικών. Αυτή θα είναι λοιπόν οι τρεις άξονες και, και δεν προτείνουν να τους αλλάξουμε. Μετά όσον αφορά το πρόγραμμα γενικότερα, ε, προσπαθούμε να υπογραμμίσουμε ότι χρειάζεται να, να δίνει έμφαση στη διαβίου μάθηση και αυτό να, να ε, ε, μεταφράζεται σε όλους τους τομείς και σε όλα τα, τα πλαίσια μέσα στα οποία μπορεί κανείς να ε, αποκτήσει γνώσεις. Υπάρχει επίσης το αίτημα να ενταθεί η συνεργασία μεταξύ τομέων. Αυτό ήταν έντονο στοιχείο του Erasmus Plus. Δημιούργησε και νέες ε, δυνατότητες συνεργασίας, για παράδειγμα μεταξύ πανεπιστημίων και οργανώσεων της νεολαίας ή αθλητικών οργανισμών. Κατά τα άλλα, οι τομεί στου οποίου απευθύνεται το Erasmus θα παραμείνουν οι ίδιοι, θα είναι και, και οι, οι εκπαιδευτικοί οργανισμοί και τα σχολεία και η τυπική εκπαίδευση και η αθλητισμό και οι οργανώσει νεολαία. Διαπιστώνουμε ότι ήταν επιτυχή η πρώτη εφαρμογή, η πρώτη προσπάθεια να εντάξουμε και τον αθλητισμό στο Εράσμο. Επέδειξε την αξία του αυτή η προσπάθεια και δημιούργησε και διάφορε πρωτοβουλίε οι οποίε καταπολεμούν του αποκλεισμού. Γι' αυτό θέλουμε να την κρατήσουμε αυτή τη δυνατότητα. Είχαμε επίσης ε, μεγάλη συμμετοχή από όλες τις χώρες Εράσμους, που δεν είναι μόνο τα 28 κράτη-μέλη. Θέλουμε να το κρατήσουμε αυτό. Όμως θέλουμε να διατηρήσουμε επίσης και την ε, δυνατότητα χωρών εταίρων που είναι ε, εκτός Ευρώπης. Όσον αφορά τον προπολογισμό, νομίζω ότι δεν είναι πάρα πολύ καλά. Ε, ε, είναι εξαιρετικό ότι θα υπάρξει διπλασιασμός του προπολογισμού, ε, γιατί γνωρίζουμε ότι πολλές από τις προτάσεις που είχαν υποβληθεί στο πρόγραμμα τελικά δεν μπορέσαμε να τις χρηματοδοτήσουμε και αυτή η αύξηση του προπολογισμού θα μας βοηθήσει να το κάνουμε στο μέλλον. Όλοι θα θέλαμε περισσότερα χρήματα, αλλά ήδη το ότι έχουμε ένα διπλασιασμό του προτινόμενου προπολογισμού είναι ένα βήμα προ τη σωστή κατεύθυνση οι προσδοκίες είναι μεγάλες. Περιμένουμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους και στην κινητικότητά τους και στην ε, διαβίου και στη γνώση. Θα πρέπει λοιπόν να προσαρμόσουμε τις διάφορες μορφές που παίρνει το πρόγραμμα για να βοηθήσουμε τους νέους, να προσπαθήσουμε το ίδιο το πρόγραμμα να καταπολεμά τους αποκλεισμούς, να γίνει πιο ε, καλό από αυτή την άποψη, και προσπαθούμε να τριπλασιάσουμε τους δικαιούχους και θα προσπαθήσω να σας εξηγήσω πώς προσπαθούμε να το κάνουμε αυτό. Δεν είναι ε, κάποιο μαγικό τρίκ, αλλά ουσιαστικά μας έχουν εμπνεύσει οι πρωτοβουλίες σε επίπεδο νεολαίας, νεολαίας που έχουμε δει ότι ήταν περισσότερο ευέλικτες και Μα το έχει δείξει και αξιολόγηση ότι χρειάζεται μεγαλύτερη ευελιξία, έτσι ώστε να μπορούν να συμμετέχουν ε, πολλών διαφορετικών ε, μορφών, ε, πολλές διαφορετικές μορφές μάθησης που μπορεί να παρακολουθεί ένας άνθρωπος. Με αυτόν τον τρόπο μειώνουμε και το μέσο κόστος, με αυτόν τον τρόπο πιστεύουμε και έχουμε υπολογίσει ότι και με το διπλασιασμό του προπολογισμού θα μπορέσουμε να τριπλασιάσουμε τους δικαιούχους. Ε, ε, και αυτός είναι ένας τρόπος για να συμμετέχουν περισσότεροι στο πρόγραμμα. Τώρα με τον διπλασιασμό του προϋπολογισμού, ε, ο διπλασιασμός μάλλον του προϋπολογισμού θα κατανεμηθεί εξίσου σε όλους τους κλάδους. Όλοι θα ωφεληθούν. Ποια είναι λοιπόν τα στοιχεία ε, της μετεξέλιξης, γιατί πράγματι δεν είναι μια επαναστατική αλλαγή, αλλά υπάρχουν κάποιες αλλαγές. Το πρώτο που σας είπα είναι ότι θα, έχουμε, θα πρέπει να φροντίσουμε το Εράσμος να απευθύνεται περισσότερο και σε ανθρώπους που έχουν λιγότερες ευκαιρίες στη ζωή τους, να καταπολεμά τους αποκλεισμούς. Ε, Ακολουθούμε επίσης κάποιες από τις συστάσεις σας. Ε, έχουμε μια νέα μορφή συνεργασίας, εταιρική συνεργασίας, στην οποία θα απευθύνεται περισσότερο σε πιο μικρές, μικρούς οργανισμούς, για παράδειγμα σχολεία, να έχουν καλύτερη πρόσβαση στο πρόγραμμα Εράσμους και αυτά. Όσον αφορά τι προσπάθειε που θα κάνουμε έτσι ώστε το πρόγραμμα καταπολεμάται τον αποκλεισμό, έχουμε μια σειρά μέτρων. Μία τις πιο, ένα από τα πιο σημαντικά είναι να προσπαθήσουμε να απευθυνθούμε περισσότερο στους τομείς εκείνους, στους κλάδους εκείνους τους οποίους δεν έχουμε την κρίσιμη μάζα, δηλαδή ε, πέρα από τα πανεπιστήμια. Οτιδήποτε εκτός από τα πανεπιστήμια. Σχολεία, μη τυπική εκπαίδευση. Και εκεί ελπίζουμε ότι οι πιο ευέλικτες μορφές συνεργασίας, οι λιγότερο βαριές, θα μας βοηθήσουν. Θα προσπαθήσουμε επίσης να αξιοποιήσουμε περισσότερο το πρόγραμμα Εράσμους για να δημοσιοποιήσουμε και να ευαισθητοποιήσουμε περισσότερο τους πολίτες όσον αφορά την Ευρώπη και την ευρωπαϊκή ταυτότητα. Ε, θα το δείτε αυτό ουσιαστικά να φαίνεται στο κεφάλαιο για τον εθελοντισμό ε, Τώρα πια έχουμε και το Ευρωπαϊκό Εθελοντικό Σώμα που μπορούμε να αξιοποιήσουμε, αλλά έχουμε επίσης και άλλες πρωτοβουλίες με τις οποίες θα προσπαθήσουμε να ενισχύσουμε τη συμμετοχή των νέων και οι οποίες ευελπιστούμε ότι θα έχουν ένα θετικό αποτέλεσμα όσον αφορά την ευρωπαϊκή ταυτότητα των νέων. Θέλουμε επίσης να απευθυνθούμε σε απόφοιτους που είχαν υποφεληθεί ε, από το Εράσμους ε, και να δημιουργήσουμε δίκτυα αξιοποιώντα τους και ε, να τους αξιοποιήσουμε στην ε, προώθηση του προγράμματος. Αναφερθήκατε κι εσεί στη σημασία που θα έχει η απλοποίηση των διαδικασιών. Συμφωνώ. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα χρειαστεί να κάνουμε σε όλα τα επίπεδα. Ήταν μία από τις προτεραιότητές μας το τρέχον πρόγραμμα. Στο, στην επόμενη εκδοχή του Εράσμου θα πρέπει να φροντίσουμε για ακόμα μεγαλύτερη απλοποίηση. Ένα στοιχείο απλοποίηση είναι αυτό που σα είπα για τι μικρή κλίμακα συνεργασία, αλλά υπάρχουν και άλλα. Θα προσπαθήσουμε να αξιοποιήσουμε περισσότερο τα εργαλεία τη πληροφορική και θα πρέπει να δούμε τι διαδικασίε τις διοικητικές για την υποβολή των αιτήσεων, έτσι ώστε να μειωθεί ο αριθμό των δικαιολογητικών και των στοιχείων που ζητούμε. Ε, βεβαίως υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί, γιατί υπάρχει ο κανονισμό για τα, ο οικονομικός για παράδειγμα, αλλά θα προσπαθήσουμε να κάνουμε όσο περισσότερη απλοποίηση μπορούμε όσον αφορά τώρα τη συνέργεια. Πράγματι, οι δράσεις μας δεν είναι αποκομμένες. Ε, υπάρχουν σημαντικοί ε, δεσμοί μεταξύ του Εράσμους και άλλων ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Για παράδειγμα, χρησιμοποιώντας κονδύλια που υπάρχουν, ε, να παραβαίνονται συμπληρωματικά προς άλλα κονδύλια που μπορεί να υπάρχουν ευρωπαϊκά. Αυτά ήθελα να σας παρουσιάσω, δεν θέλω να μακρηγορήσω. Μπορώ να απαντήσω και σε ερωτήσει. Ελπίζω να σας έδωσα τα κύρια στοιχεία της νέας μας πρότασης. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Τριπλασιασμός ε, των ε, συμμετεχόντων. Με διπλασιασμό όμως των κονδυλίων. Ε, πώς θα το κάνουμε αυτό το μαγικό. Είπατε ότι θα πρέπει να υπάρχουν πιο πολλές εικονικές ε, επαφές. Τελική ανάλυση, δηλαδή αυτό τι σημαίνει, ότι αυτοί που έχουν χρήματα θα έχουν ε, πραγματικό ταξίδι και οι υπόλοιποι που δεν έχουν χρήματα θα έχουν μόνο εικονική επαφή με τα πανεπιστήμια. Να περάσουμε πρώτα στους εισηγητές και στον εισηγητή και στους κοιόδες εισηγητές. Να ακολουθήσουμε τη διαδικασία ping-pong. Ο συνάδελφο Φέρο, ο οποίο είναι και εισηγητή, είναι ο πρώτο που θα πάρει το λόγο για πέντε λεπτά. Κατά το όριο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητοί σκιώδες εισηγητέ, σας ευχαριστώ που μου κάνετε την τιμή να με διορίζετε εισηγητή σε ό,τι αφορά τα θέματα αυτά, είναι γνωστό ότι στις 13 Μαΐου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταθέσει μια επιτροπή για διπλασιασμό των κονδυλίων για το επόμενο πολιτικό δημοσιονομικό πλαίσιο. Μετά το Brexit θα πρέπει να δούμε και μείωση των μέσων σε ό,τι αφορά την πολιτική συνοχή, σύμφωνα με την πρόσθεση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο επόμενο πολιτικό δημοσιονομικό πλαίσιο και θα πρέπει, φαντάζομαι, εν ώψη και των αλλαγών αυτών, να θεωρήσουμε επιτυχία το διπλασιασμό των μέσων αυτών. Μιλάμε λοιπόν για 15 δις. Θα υπάρχουν λοιπόν 30 δις και θα πρέπει να συνυπολογιστεί και ο πληθωρισμός. Από την άλλη, έχουμε και νέες πρωτοβουλίες ε, προς χρηματοδότηση ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, κέντρα σε διάφορα προγράμματα όπως το Discovery EU. Σε τελική ανάλυση θεωρώ δηλαδή ότι θα είναι πιο περιορισμένοι οι πόροι από ό,τι αναμένουμε. Θα πρέπει να γίνει η κατανομή των κονδυλίων και πιστεύω ότι η προτεραιότητα της Επιτροπής Πολιτισμού και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα πρέπει να είναι να τηρήσουμε αυτά που είχαμε ζητήσει για το πολιτισμικό πλαίσιο. στα πλαίσια του τριπλασιασμού που είχαμε ζητήσει. Μιλάμε για μία από τις πιο σημαντικές, ε, ένα από τα πιο σημαντικά καθήκοντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, σε ό,τι αφορά την κατάρτιση, τη συνοχή και θα ήθελα να κοιτάξουμε τις ε, προτάσεις από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το νέο πρόγραμμα λοιπόν θα ονομάζεται πλέον Erasmus Plus. Θα φέρει αυτό το θετικό πρόσημο, ήταν 7ο έτος για το πρόγραμμα αυτό. Και χαίρομαι που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν τροποποίησε το βασικό οικοδόμημα του προγράμματος. Εξακολουθούν να υπάρχουν ε, τρία προγράμματα για την κινητικότητα των ατόμων, για τη συνεργασία μεταξύ των οργανώσεων και για την ανάπτυξη της πολιτικής ε, κατάρτισης. Όπως σας είπα, έχουμε και νέες πρωτοβουλίες, οι οποίες ε, θεωρώ ότι θα διαδοθούν ταχύτατα και θα συνδράμουν στη διατήρηση και της ευρωπαϊκής ταυτότητας αλλά και της ε, ευρωπαϊκής κληρονομιάς. Θεωρώ ότι όλα αυτά λοιπόν περιλαμβάνονται στα διάφορα προγράμματα όπως για παράδειγμα το Discovery EU. Καλώς ορίζω το γεγονό ότι υπάρχουν και άλλες δύο πρωτοβουλίες για τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, τα κέντρα για την επαγγελματική κατάρτιση και την επαγγελματική πιστοποίηση. Τα κέντρα λοιπόν αυτά είναι στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής προσοχής τα τελευταία χρόνια και σκοπός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι να αυξήσουν να αυξηθούν, να διπλασιαστούν και τα κονδύλια και ο αριθμό των συμμετεχόντων. Και αυτό λοιπόν το καλωσορίζουμε. Δεν είναι μόνο απαραίτητο να συμπεριληφθούν οι πανεπιστημιακοί φοιτητέ, αλλά και οι μαθητευόμενοι, οι μαθητές, οι δάσκαλοι, οι εκπαιδευτές, ε, Και θα ήθελα να αναφέρω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο... στην πρόταση της δεν, αναφέρει τον κοινοβουλευτικό έλεγχο. Είναι σημαντικό λοιπόν να τονίζουμε την τύχη αυτή του προγράμματος. Νομίζω ότι μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα βρούμε λύσεις για το πώς μπορούμε να συμπεριλάβουμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στον τρόπο λειτουργία του προγράμματος. Σημαντικό είναι επίση το πρόγραμμα αυτό να ισχύει και για τα άτομα τα οποία βρίσκονται στο περιθώριο τη κοινωνία. Είναι θετικό ότι θέλουμε να απλοποιήσουμε τι διαδικασίε, να διπλασιάσουμε τα κονδύλια, να μειώσουμε τα γραφειοκρατικά εμπόδια και από ό,τι ακούσαμε σήμερα γίνονται συγκεκριμένα βήματα προ την κατεύθυνση αυτή για την απλοποίηση. Αλλά σε πολλές περιπτώσεις ε, δεν επαρκούν όλα αυτά και γι' αυτό συμφωνώ με την τελευταία σκέψη που εκφράστηκε. Συμφωνώ με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι θα πρέπει το συντομότερο δυνατόν να βρούμε μια συμφωνία για το επόμενο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο κατά προτίμηση μέσα στο 2019, γιατί αν υπάρξει καθυστέρηση, ενδεχομένω ε, να υπάρχουν συνέπειε σημαντικέ για, για το πρώτο έτος του επόμενου πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου. Θα κάνω λοιπόν ό,τι περνάει από το χέρι μου για να επιταχύνω τη διαδικασία αυτή. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και του σκιώδε εισηγητέ και τα μέλη τη Επιτροπή Πολιτισμού. Με τη συνεργασία μα θεωρώ ότι θα πετύχουμε το στόχο μα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, Λεκύη Πρόεδρο. Και δεν ξέρω αν θα θέλετε να πάρετε το λόγο για να απαντήσετε. Μήπω να ακούσουμε πρώτα και του υπόλοιπου συναδέλφου. Μάλιστα. Αν υπάρχουν λοιπόν συγκεκριμένε ερωτήσει από πλευρά σα να τις απευθύνουμε είτε στου εμπειρογνώμονε, είτε προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ξεκαθαρίσετε στις παρεμβάσει σα, γιατί άλλο θα θεωρήσω ότι έχετε προβεί σε δηλώσει και σε ανταλλαγή απόψεων. Και στην περίπτωση αυτή θα δώσουμε το λόγο στο τέλο προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στους εμπειρογνώμονε. Συνάδελφο Λιμπάτσκα, σα παρακαλώ μην υπερβείτε τα τρία λεπτά όμω. Ευχαριστώ. Το Εράσμος είναι πολύ γνωστό, αναγνωρίζεται ότι είναι αποτελεσματικό και αυτό το ξέρουμε όλοι μας. Συχνά τονίζεται ότι διπλασιάστηκαν τα κονδύλια για το Εράσμους. Χαιρόμαστε γι' αυτό. Αλλά ας σκεφτείτε τα πολλαπλά καθήκοντα του Εράσμους, παρότι έχουμε διπλασιάσει τον προϋπολογισμό, δεν φτάνουν τα λεφτά. Έχουμε τριπλασιασμό του αριθμού των συμμετεχόντων. Ε, Ευρωπαϊκός χώρος εκπαίδευσης, νέα πρόκληση. Ευρωπαϊκά, δίκτυα μάλλον Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων, νέα πρόκληση. Ε, η νέα πρόκληση είναι επίσης ε, οι μετακινούμενοι καθηγητές ανά την Ευρώπη. Ο διπλασιασμός λοιπόν των ε, πόρων δεν αρκεί. Είναι όλο και λιγότερος όταν βλέπετε πόσα πολλά πράγματα καλύπτει το Εράσμους. Επομένως, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να εξασφαλίσουμε αύξηση και της χρηματοδότησης του Εράσμους. Δεύτερον, σε κάθε αναθεώρηση, σε κάθε επανεξέταση του προγράμματος, μας απασχολεί ο μεγάλος ε, βαθμός επιτυχίας, δηλαδή ο πολλαπλός αριθμός χρηματοδότησης σχεδίων. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρξει επιπλέον χρηματοδότηση αυτών των προγραμμάτων από το... και να χρηματοδοτηθούν από τον ορίζοντα 2020. Μήπως θα μπορούσαμε να έχουμε αυτή την ε, ευελιξία. Μήπως θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε καλύτερα το εράσμους και το ορίζοντα 2020. Επίσης, τα ποσά των επιχορηγήσεων που δίνεται, να τα προσαρμόσετε στο κόστος ζωής της κάθε χώρας. Επίσης, τι θα γίνει με την υποστήριξη των ε, εθνικών οργανισμών, ε, εκείνων που δυσκολεύονται. Επίσης, μπορείτε να μιλήσετε λιγάκι περισσότερο για την πρωτοβουλία ανακάλυψη της Ευρώπης, γιατί το βασικό μας θέμα είναι η επικοινωνία. Το να του δώσουμε ένα εισιτήριο κανενό δεν σημαίνει ότι θα μπορέσει να πληρώσει για να επισκεφθεί την Ευρώπη. Είπατε επίση ότι υπάρχει μια ιδέα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την καλύτερη συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Μπορείτε να μα πείτε περισσότερα και λίγα περισσότερα πράγματα θα ήθελα να ακούσω για την, ε, τις συνέργειες ανάμεσα στο Εράσμος και τον Ορίζοντα 2020. Σύντομα, αν μπορείτε, παρακαλώ. Θα προσπαθήσω, λέει εκπρόσωπος Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Να σας πω κάποια πράγματα τώρα. Χρήσιμες ήταν οι ερωτήσεις που ακούστηκαν. Για το ποσοστό επιτυχίας ε, και, τα, και την αύξηση του προϋπολογισμού. Ξέρουμε ότι υπάρχει απογοήτευση στον κλάδο από κάποιους, γιατί δεν υπάρχουν αρκετά κονδύλια. Στο σχεδιασμό, λοιπόν, θα δείτε ότι Προσπαθούμε να προτείνουμε αύξηση για τις διάφορες βασικές ε, δράσεις σε διάφορους τομείς και θα δείτε ότι θα υπάρξει βελτίωση σε αυτό το επίπεδο. Φυσικά δεν θα υπάρξει ποτέ βαθμός ε, επιτυχίας των σχεδίων 100%. Υπάρχει ένα ανώτατο όριο, όμως θα χρηματοδοτούνται περισσότερα προγράμματα σήμερα. Στον τομέα της νεολαίας είχαμε το χαμηλότερο βαθμό επιτυχίας. Γι' αυτό το κεφάλαιο για την νεολαία το διπλασιάσαμε και αυτό είναι σημαντικό μήνυμα που θέλουμε να στείλουμε στην νεολαία. Ε, θα προσπαθήσουμε να τονώσουμε την, ε, τις εταιρικές σχέσεις και κτλ. Σε αυτόν τον τομέα. Για τη σχέση με τα άλλα προγράμματα. Πολύ σημαντικό σημείο. Να σας πω δύο λόγια γι' αυτό. Ε, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Plus ε, είναι και αυτό παράλληλα στο τραπέζι. Ε, και έχουμε συνεργαστεί με τους συναδέλφους στη Γενική Διεύθυνση Απασχόληση. Έχουμε δύο συγκεκριμένε ιδέε για το πώ θα βελτιώσουμε τι συνέργειε ανάμεσα στα δύο. Καταρχά το ένα συνδέεται με το βαθμό επιτυχία των ε, προγραμμάτων. Δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε τον ίδιο μηχανισμό με τον ορίζοντα, αλλά θέλουμε προγράμματα τα οποία δεν έχουν επιτύχει πλήρως το Erasmus Plus να έχουν τη δυνατότητα να συνεχιστούν ε, στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου Plus. Ε, θα δούμε τους τρόπους, αλλά αυτή είναι μια σκέψη. Από την άλλη, υπάρχουν καλά και καινοτόμα προγράμματα που έχουν επιτύχει και θεωρούμε ότι είναι καλές πρακτικές, είναι υπερεθνικά, διεθνικά προγράμματα και πιστεύουμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο μπορεί να τα αναβαθμίσει σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο. Αυτές είναι οι ιδέες που επεξεργαζόμαστε αυτή τη στιγμή. Προσπαθούμε να βρούμε τους τρόπους. Είναι σημαντική η σχέση επίσης με το ε, Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο για να συμπληρώνει τα κονδύλια. Δηλαδή, σε ένα πρόγραμμα, εάν το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο είναι σημαντικό για αυτή την περιοχή ή για αυτή τη χώρα και υπάρχει προτεραιότητα για μια συγκεκριμένη ομάδα, θα πρέπει να συμπληρώνονται τα κονδύλια του Εράσμου από το ESF+, από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Plus δηλαδή. Θα δούμε πώς θα λειτουργήσει αυτό, αλλά αυτή είναι η ιδέα που έχουμε σκεφτεί ε, προετοιμάζοντας την πρόταση για τα δύο προγράμματα. Υπάρχουν πολλοί σύνδεσμοι με τον ορίζοντα. Ε, η έρευνα ε, στα, των Ευρωπαϊκών ε, Πανεπιστημίων μπορεί να χρηματοδοτηθεί μέσω του ορίζοντα, Φερρυπίν. Σε ό,τι αφορά τις επιχορηγήσεις που αναφέρατε, είναι σημαντικό θέμα αυτό. Θα πρέπει να κάνουμε κάποιες μελέτες ε, και να καταλάβουμε πλήρως ποια είναι η κατάσταση, γιατί αλλάζει συνέχεια, αλλά η κατάσταση των δανείων και των επιχορηγήσεων πρέπει να ευθυγραμμιστεί με την πραγματικότητα, με το ποιο είναι το πραγματικό κόστος. Θα αναθεωρήσουμε το σύστημα αυτό λοιπόν των επιχορηγήσεων και δανείων και αν χρειάζεται θα το αλλάξουμε. Η ιδέα πάντως είναι να δίνουμε επιπλέον επιχορηγήσεις για ανθρώπους με λιγότερες ευκαιρίες όταν χρειάζεται. Ε, θέλουμε λοιπόν να δούμε ποιες είναι οι εταιρικέ σχέσεις και να δώσουμε κίνητρα μέσω του συστήματος ε, των επιχορηγήσεων. Σας ευχαριστώ. Επόμενος είναι η συνάδελφος Μαρίτερα Στοιχειομένης για τρία λεπτά. Ah, ευχαριστώ για την παρουσίαση αυτής της μελέτης που ήταν ενδιαφέρουσα και εγώ έχω μια-δυο ερωτήσεις. Σε αυτή την ε, ανταλλαγή απόψεων Πρέπει να σας πω ότι το πρόγραμμα ΕΡΑΣΜΟΣ είναι το, το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δίνει αυτή την αίσθηση ότι η Ευρώπη είναι η γη όλων μας. Είναι για τους νέους, είναι για την εκπαίδευση, για τη συνεργασία και την κινητικότητα μεταξύ των κρατών μελών. Κάτι που με ενδιαφέρει όλος ιδιαίτερος είναι οι δυνατότητες που έχει για ανταλλαγές με τις συνδεδεμένες χώρες. Είμαι πρόεδρος της αντιπροσωπείας για το Μαγκρέμπ. Και υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορούμε να κάνουμε στη Βόρεια Αφρική. Τι μέσα έχουμε για να κάνουμε κάποια πράγματα και από την άλλη όχθη της Μεσογείου. Επίσης, μια άλλη ερώτηση που θέλω να σας κάνω ότι εμείς είχαμε κάποιες ιδέες για τα χρήματα. Το είπε και η Πέτρα, δεν είμαστε απόλυτα ευχαριστημένοι για το θέμα των, της χρηματοδότησης. Θα ήθελα να μου πείτε δύο λόγια για την μελλοντική σχέση ε, του Ηνωμένου Βασιλείου με το Εράσμους. Γιατί ξέρατε ότι το 2016 26.800 Ευρωπαίοι συμμετείχαν ε, στο στις αυτές τις ανταλλαγές μέσω του Εράσμους και οι 1500 ήταν από το Ηνωμένο Βασίλειο. Από το Μάρτιο του 2019, τι θα γίνει με αυτούς τους μαθητές, με αυτούς τους φοιτητές, τους σπουδαστές κτλ. Και μια άλλη ερώτηση. Υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός Ευρωπαίων ε, ε φοιτητών που ενδιαφέρονται για επιστημονική καριέρα. Επομένως είναι σημαντικό η Ευρώπη να προχωρήσει και να ανταγωνίζεται για την πρόθεση της ευρωπαϊκής επιστήμης. Τι μέσα θα πάρει η Κομισιόν μέσω του Εράσμους για να προωθήσει τις ανταλλαγές για την, στον τομέα της επιστήμης, τεχνολογίας, στη μηχανική και στα μαθηματικά όλος ιδιαίτερος. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Η επόμενη μιλήτρια για να απαντήσει η κυρία Έριξον. Σας ευχαριστώ πολύ. Πολλά καλά στοιχεία μας επισημάνατε. Σας ευχαριστώ. Και θα προσπαθήσω να απαντήσω σε τρία εξ αυτών. Το διεθνέ ε, θέμα, το θέμα του Ηνωμένου Βασιλείου και το θέμα της επιστήμης. Ε, σε ό,τι αφορά το διεθνές επίπεδο ήταν πολύ καλή η συνεργασία με τις χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρίως με τις γειτονικές χώρες και προφανώς αυτό θα συνεχιστεί. Ήταν πολύ καλή συνεργασία στον τομέα της νεολαίας, στον τομέα της ανατολής εκπαίδευση. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν να το επεκτείνουμε αυτό και σε νέου τομεί. Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Υπάρχει λοιπόν αυτή η, αυτό το αίτημα και από δική σα πλευρά. Με το πρόγραμμα Εράσμου, λοιπόν θα πρέπει να δούμε ότι με το προπολογισμό μα δεν μπορούμε να τα πετύχουμε όλα. Προφανώ. το Εράσμου μπορεί να επιδιώξει του τους μα, εσωτερικού ευρωπαϊκού στόχου. Θα πρέπει να δούμε και τα εξωτερικά εργαλεία τα οποία υποστηρίζουν τις δραστηριότητε, για παράδειγμα την οικοδόμηση δυναμικού στους τομείς αυτούς. Εκεί έχουμε και την χρηματοδότηση των εξωτερικών εργαλείων. Άρα και στο Erasmus Plus έχουμε κάποιες δραστηριότητες όπου μπορούμε να συνδυάσουμε τους στόχους αυτούς. Και αυτό προβλέπουμε και για το μέλλον. για το Ηνωμένο Βασίλειο. Δυστυχώς ε, δεν βλέπω να μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα, γιατί πολύ απλά δεν ξέρουμε πού βρισκόμαστε, είμαστε στα χέρια. Μια ε, μελλοντική συμφωνία το καθεστώ του Ηνωμένου Βασιλείου δεν είναι σαφέ. Μετά το Brexit δεν είναι σαφέ. Πολύ απλά δεν ξέρουμε. Αυτό είναι το... αυτό που έχω να πω για την ερώτησή σα. Για την επιστημονική πλευρά δεν το ανέφερε αυτό. Είναι μια μεταξέλιξη, είναι μια νέα ένα νέο τομέα όπου θέλουμε να προωθήσουμε την κινητικότητα σε στρατηγικού ε, τομεί, για παράδειγμα κινητικότητα στο STEM, STEAM, σε ό,τι αφορά την αλλαγή του κλίματος, σε ό,τι αφορά την ενεργειακή αποδοτικότητα, τεχνητή νοημοσύνη. Όλοι αυτοί οι τομείς, ε, οι μελλοντοστραφείς, αν θέλετε, δίνουν μια κάποια προπτική. Είναι ειδικέ λοιπόν αυτές τις δραστηριότητε τις οποίες θέλουμε να ενθαρρύνουμε στα πλαίσια τη κινητικότητα και τη ανώτατη εκπαίδευση, όχι όμω απαραίτητα μόνο σε αυτού του τομεί. Ευχαριστώ. Μάλιστα, λέει η πρόεδρο. Η συνάδελφο, η κυρία Εύανση, για τρία λεπτά, παρακαλώ. Ευχαριστώ, πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και για την πολύ ενδιαφέρουσα και θετική παρουσίαση και καταρχάς θα ήθελα να συμφωνήσω με τα σχόλια των συναντέλφων ε, σε ό,τι αφορά την ε, χρηματοδότηση και θα υποστηρίξω και εγώ τον τριπλασιασμό των πόρων. Θα ήθελα επίσης να αναφερθώ στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου. Λέτε δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Αλλά Βεβαίω η Ουελία, την οποία εγώ εκπροσωπώ έχει την επιθυμία και να παραμείνει στο Εράσμους και θα το προσπαθήσουμε οποιοδήποτε και είναι το αποτέλεσμα και οποιοδήποτε θέση ε, τηρήσει η Βρετανική κυβέρνηση. Η Ουελία τουλάχιστον θα προσπαθήσει να επανενταχθεί, να ενταχθεί, να παραμείνει γιατί έχουμε διαπιστώσει πόσο μεγάλη είναι η ισχύ του Εράσμους, πόσο μπορεί να μετασχηματίζει τα πράγματα και πόσο ε, σημαντική ε, ε, πόσο σημαντική είναι η ευρωπαϊκή συνεργασία και πώς αυτό το επιδεικνύει το Εράσμος, καταδεικνύει το Εράσμος. Θα ήθελα να σας κάνω μια συγκεκριμένη ερώτηση όσον αφορά την δυνατότητα εγγύησης των φοιτητικών δανείων. Είναι κάτι το οποίο ανέφερε η κυρία Φαντερκράφ ότι τα αποτελέσματα εδώ δεν ήταν τα αναμενόμενα. Θα ήθελα να μου πείτε ποια είναι κατά την άποψή σας οι λόγοι. Από την εμπειρία τη δική μου από τα πανεπιστήμια στην Ουαλία, είναι ότι συνήθως οι φοιτητές οι οποίοι ζητούν ανταλλαγές εράσμους είναι φοιτητές ε, γλωσσών. Και ε, σπανιότερα έχουμε αιτήσει για ανταλλαγές εράσμους σε άλλους τομείς θα ήθελα να μου πείτε αν αυτό είναι ένα έβριμα που το επιβεβαιώνετε κι εσείς, το είδατε στη διαβούλευση και αν ναι, εάν έχετε σκεφτεί κάποιες λύσεις ε, για να το αντιμετωπίσουμε. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω το λόγο στην κυρία Φαντεγκράφ πρώτα για να απαντήσει σε αυτή την ερώτηση. Γιατί είναι έτσι τα πράγματα γιατί το, τα φοιτητικά δάνεια, η γεωδοσία τους δεν λειτουργεί όπως θα θέλαμε. Κυρία Φαντεγκράφ, το σύστημα γεωδοσίας των φοιτητικών δανείων είναι ένα σύστημα που πράγματι, όπως σας είπα, είχε αποτελέσματα ανάμεικτα. Πέντε τράπεζες έχουν συμμετάσχει στο πρόγραμμα, επομένως ήδη είναι μικρός ο αριθμός των τραπεζών που μπορούν να βοηθήσουν. Πέραν αυτού πιστεύω ότι δεν έχουν υπάρξει κίνητρα για να αυξηθεί ο αριθμό των τραπεζών που θα συμμετείχαν, γιατί σε μεγάλο βαθμό τα κράτη-μέλη έχουν εθνικά συστήματα υποστήριξης και επίσης είναι και μικρός ο αριθμός των δικαιούχων των παιδιών που θέλουν να συμμετάσχουν. Ίσως να μην είναι γνωστά, ε, γνωστές αυτές οι δυνατότητες. Εμείς ε, σταθήκαμε πολύ περισσότερο στο επίπεδο των δικαιούχων για να ακούσουμε τη δικιά τους εμπειρία και διαπιστώσαμε ότι πολύ λίγοι από τους δικαιούχους γνώριζαν ότι υπήρχαν, είχε αυτή η δυνατότητα. Επομένως αυτά τα τρία στοιχεία είναι πιστεύω που εξηγούν σε μεγάλο βαθμό το κατάσταση με αυτό το σύστημα. Σας ευχαριστούμε πολύ, λέει η Πρόεδρος. Πριν να δώσω πάλι λόγο στην κυρία Ρίξον... Θα ήθελα να καλωσορίσω 35 επισκέπτες από τη Βουλγαρία που βρίσκονται ε, στο πίσω μέρος της αίθουσας μετά από πρόσκληση του συναδέλφου κυρίου Νέκοφ. Καλωσορίσατε. Ελπίζω να ε, σας φανεί ενδιαφέρουσα η συζήτησή μας σήμερα το πρωί. Κυρία Άριξον. Ευχαριστώ. Για τα αυτιλικά δάνεια. Πράγματι, ε, από τη δημόσια διαβούλευση της Επιτροπής κάτι αντίστοιχο διαπιστώσαμε και εμείς το βλέπουμε και από την εφαρμογή του προγράμματος φάνηκε ότι ήταν δύσκολο ε, να ξεκινήσει αυτό το σύστημα να λειτουργεί και ε, εμείς αντιλαμβανόμαστε ότι δεν ήταν ελκυστικό το πρόγραμμα αυτό για το, τις, χρημα, τις οργανώσεις χρηματοδότησης, τους οργανισμούς χρηματοδότησης πέραν από αυτούς τους 5-6 που συμμετείχαν, ήταν δύσκολο, διαπιστώσαμε ήταν δύσκολο να, να, να πείσουμε ε, τις τράπεζες και άλλους τέτοιους οργανισμούς να συμμετάσχουν. Αυτό έχει σχέση με την κατάσταση της χρηματοοικονομικής ε, αγοράς. Ε, γι' αυτόν τον λόγο αποφασίσαμε να το καταργήσουμε. δεν θα το δείτε στη νέα πρόταση για το Εράσμους. ίσως να συνεχίζουν να υπάρχει η ανάγκη για ένα τέτοιο σύστημα σε κάποιες περιπτώσεις. Θα μπορούσε κανείς να αξιοποιήσει περισσότερο το σύστημα InvestEU, αυτά τα ευρωπαϊκά προγράμματα, υπάρχει δυνατότητα από εκεί. Βέβαια, το πρόγραμμα επενδύοντα στην Ευρώπη δεν αφορά μόνο στην κατάρτιση και την εκπαίδευση, είναι πολύ ευρύτερο, αλλά θα μπορούσε κανείς να αξιοποιήσει αυτή τη δυνατότητα που προκύπτει από έναν ξεχωριστό, έναν διαφορετικό κανονισμό. Είναι ενδιαφέρον αυτό που μου λέτε για τους ε, φοιτητέ που σπουδάζουν ε, γλώσσες. Γνωρίζουμε ότι η γνώση μιας ξένης γλώσσας πολύ συχνά είναι φραγμός στο να προσπαθήσει κανείς να πετύχει ένα πρόγραμμα ανταλλαγή. Γι' αυτό το ε, χτες κιόλας κάναμε κάποιες προτάσεις ως Ευρωπαϊκή ε, Επιτροπή για την ενίσχυση της γλωσσομάθειας. Ε, αυτό βέβαια θα αλλάξει από τη μια μέρα στην άλλη. Πρέπει να ενθαρρύνει κανείς την εκμάθηση ξένων γλωσσών από την ε, παιδική ηλικία. Έχουμε κάποιες προτάσεις σε αυτή τη σύσταση και ελπίζουμε τα κράτη-μέλη να τις ακολουθήσουν ελπίζουμε ότι με αυτόν τον τρόπο θα βρεθούν περισσότεροι φοιτητέ που θα τολμήσουν να πάνε σε μια χώρα του εξωτερικού να σπουδάσουν ένα εξάμεινο ή περισσότερο. Ε, Βεβαίω υπάρχουν και άλλε δυνατότητε. Μπορεί να υπάρχει ένα πρόγραμμα προπαρασκευαστικό ή ένα πρόγραμμα βελτίωση τη ξένη γλώσσα όταν κανεί βρίσκεται στο Εράσμο, αλλά πρέπει να ξεκινάει ήδη με καλέ βάσει. Σα ευχαριστώ και θυμάμαι πολύ καλά τη συζήτηση που είχε γίνει τότε για τα δάνεια προς τους φοιτητές ήταν πραγματικά κάτι το οποίο ήταν αμφιλεγόμενο και στα πλαίσια της Επιτροπής μας. Δεν ήμασταν βέβαιοι κατά πόσον όντως επρόκειτο για ένα μέσο το οποίο θα είχε αποτέλεσμα ή το οποίο ενδεχομένω να ήταν καλύτερα να το αφήσουμε. Τότε λοιπόν είχαμε πει ότι θα το δοκιμούσαμε, το δοκιμάζαμε και ότι θα βλέπαμε, εν πάση περιπτώσει, αν ε, λειτουργούσε ή όχι. Αυτή λοιπόν ε, είναι η ιδέα καθοδήγηση από την ε, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ναι, για να μην υπάρχει ουσιαστικά τόσο μεγάλη συμμετοχή των ιδιωτικών τραπεζών αλλά πιο πολύ από την ΕΤΕΠ. Να πούμε ότι υπάρχει τουλάχιστον σε κάποιου τομεί η δυνατότητα αυτή και αν τα χρήματα αυτά δεν χρησιμοποιηθούν τουλάχιστον δεν θα πάνε και χαμένα. Ολοκληρώσαμε λοιπόν τον γύρο των σκιωδών εισηγητών. Και θα περάσουμε τώρα στα υπόλοιπα μέλη που έχουν ζητήσει το λόγο από πλευρά τη Ευρωπαϊκή της Επιτροπής μας. Δύο λεπτά παρακαλώ ο καθένας. Έχουμε άλλη μια ωρίτσα. Αν θέλετε να ζητήσετε εκ νέου το λόγο στη συνέχεια. Να ξεκινήσουμε με την κυρία Σόιντροβα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Οι συνάδελφοι Ευχαριστώ και του συναδέλφου. Ξέρω ότι η, η πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, έλαβε υπόψη αυτά που ε, εγκρίθηκαν και αυτά που δεν εγκρίθηκαν θα συνεχίζουν. Υπάρχουν κάποια καινούργια πολιτικά προγράμματα. Για το Discovery EU, για παράδειγμα, για τα νέα πολιτικά αυτά προγράμματα, έχω κάποιε ερωτήσει να κάνω. Αυτό το Discovery EU, πώ θα λειτουργήσει, πώ θα το εξηγήσουμε στα σχολεία. τα σχολεία μας δηλώνουν ότι υπάρχει ένας ανταγωνισμός σε ό,τι αφορά τα project, σε ό,τι αφορά τα έργα και τώρα δίνουμε ένα πρόγραμμα το οποίο δεν έχει ανταγωνισμό, δεν έχει ε, οδικό χάρτη. Ύστερα, το θέμα της κινητικότητας. Σε επίπεδο του Citizens for EU. Νομίζω ότι τέριαζε καλύτερα το θέμα αυτό. Νομίζω ότι αυτό πολύ απλά αφαιρεί πόρους από την εκπαίδευση από το εράσμος. Νομίζω ότι τα πολιτικά προγράμματα λοιπόν θα δείξουν προς τα που οδεύουμε το δεύτερο θέμα των Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων. Και εδώ έχω μια ερώτηση να κάνω. Πιστεύω ότι σήμερα ήδη το θέμα της αριστείας είναι ιδιαίτερα σημαντικό και συμφωνώ να υπάρξει μια ευρωπαϊκή, αν θέλετε, επισήμανση, ένα ευρωπαϊκό σήμα για τα πανεπιστήμια. Αλλά έχω επιβολή για το πώς θα λειτουργήσει το θέμα. Και νομίζω ότι συνδέεται αυτό φυσικά και με τον πρόεδρο Μακρόν, αλλά να μην τα επικεντρώνουμε όλα αυτά σε πολιτικό επίπεδο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, λέει η πρόεδρο, σε, ό,τι αφορά το ερώτημα για το Discover EU. Αυτό δεν ορίζεται καν στο κείμενο, αναφέρεται, καν, αναφέρεται ως όρος. Το τι θα περιλαμβάνει στην τελική ανάλυση θα το αφήσουμε στην διακριτική ευχαίρεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ερωτηματικό. Κύριε Έριξον. E το ανακαλύπτοντας την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι διτό. Πρέπει να δούμε τι κάνουμε τώρα κατόπιν ετήσεως και του Κοινοβουλίου. Είναι να εφαρμόσουμε το Discovery ως προπαρασκευαστική δράση. Ε, ζητήθηκε να, εφαρμόσουμε, να το εφαρμόσουμε το συντομότερο δυνατόν, μάλιστα. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε. Ε, για να επιτρέψουμε τους, στους πρώτους νέους να ταξέψουν φέτος το καλοκαίρι σε μια πρώτη πιλωτική φάση. Φυσικά πρέπει να γίνουν κάποιες επιλογές, ε, γίνεται κάποιος ανταγωνισμός, ε, αλλά θα είναι μια πιλωτική φάση και αυτό είναι θετικό. το feedback που παίρνουμε είναι πολύ ενθαρρυντικό. Ε, υπόσχεται πολλά αυτό το project. Στο μέλλον ε, το γεγονό ότι αυτό, σε αυτή τη φάση είναι προπαρασκευαστική δράση δεν έχει καμία σχέση με το Εράσμους. Πρέπει να την κάνουμε αυτή τη διάκριση. Η πρότασή μας τώρα είναι να μάθουμε από αυτή την πιλωτική φάση και αν θα υπάρξει τώρα μια νέα του χρόνου θα μάθουμε πάλι ακόμα περισσότερο και θα προτείνουμε μια καλή πρόταση για μια καλή πρωτοβουλία από το 2021 πια. Ε, το μελλοντικό Discovery, Discovery U δεν θα εφαρμοστεί όπως σήμερα. Ε, αν είναι τμήμα του Εράσμους, θα πρέπει να εντάσσεται στους συνολικούς στόχους του Εράσμους. Θα πρέπει να έχουμε ένα στόχο μαθησιακό και εκπαιδευτικό, πολύ έντονο. Τώρα έχουμε το πλαίσιο, έχουμε προτείνει το πλαίσιο, θα πρέπει να μάθουμε και θα πρέπει, και αυτό που συζητάμε τώρα, είναι να προετοιμάσουμε την εφαρμογή. Το πώς θα εφαρμόσουμε αυτή την πρωτοβουλία είναι τμήμα αυτού του προβληματισμού που θα την κάνουμε μαζί με εσά. Είναι σημαντικό να μην ξεχνάμε ότι θέλουμε να έχουμε μια ισχυρή μαθησιακή διάσταση στο μέλλον και το Discover You πρέπει να, έχουμε, να έχει σχέση με την συγκεκριμένη κοινότητα ε, με την περιοχή. Θα πρέπει να εμπλέξουμε και οργανώσεις νεολαίας και άλλες οργανώσεις για να βρουν τους ανθρώπους που δεν έχουν κατανάγκη ανάγκη τις δυνατότητε να ταξιδέψουν από μόνοι τους. Αυτή είναι η ιδέα που έχουμε στο μέλλον. Ευχαριστώ. Όταν συζητήσουμε το Erasmus Plus και το σχετικό κανονισμό, θα πρέπει να σκεφτούμε και εντός του Κοινοβουλίου πώς το Discovery U, το ανακαλύπτοντας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μπορεί να γίνει πολύ πιο συγκεκριμένο και να συνδεθεί με τους στόχους του Εράσμους, ούτως ώστε να έχουμε και τη διάσταση της κινητικότητας και τη διάσταση της ε, εκπαίδευσης. Το θέμα δεν είναι να είσαι τουρίστα στην Ευρώπη. Ε, το ταξίδι έχει να κάνει και με την επικοινωνία και με την εκπαίδευση. Είτε τυπική είτε μη τυπική. Θα πρέπει λοιπόν να το συζητήσουμε αυτό το θέμα. Η κυρία Χέλγκα Τρίπελ είναι η επόμενη. Ευχαριστώ, Πέτρα. Θα ήθελα να πω από την αρχή ότι για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην έχουμε απλώς ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για φοιτητέ. Είναι πολύ πιο ευρύ το θέμα. Ε, νέοι άνθρωποι, άντρες και γυναίκες, ε, και να ξεπερνάμε και την διάσταση της Ευρώπης, να αποκτήσει μια διεθνή διάσταση. Να μην το ξεχνάμε αυτό. Υπάρχει και μια κοινωνική βέβαια διάσταση. Δεν θέλουμε απλώς να φτώσουμε εκείνους που ξεκίνησαν καλά στη ζωή και άνετα. Θέλουμε να φτάσουμε και σε εκείνους που δυσκολεύτηκαν περισσότερο να αποκτήσουν τέτοιες ευκαιρίες. Ε, και αυτοί οι άλλοι άνθρωποι, οι πιο μειονεκτούντες θα πρέπει να υποφεληθούν. Τώρα, για τις κατεξιοδότηση ή εκτελεστικές πράξεις. Πέτρα, σε υποστηρίζω. Εμείς ως Κοινοβούλιο θα περάσουμε σε μια πολύ δύσκολη διαπραγμάτευση για τα δικαιώματα του Κοινοβουλίου σε ό,τι αφορά την εφαρμογή και εκτέλεση του προγράμματος. Θέλουμε να παίξουμε ένα ρόλο εδώ. Δεν μπορούμε να δεχτούμε η Κομισιόν να αποφασίζει με μη διαφωνείς ε, τρόπους για αυτές τις πολιτικές. Θα γίνει σκληρή διαπραγμάτευση και πρέπει να συμμετάσχουμε. Τώρα για τον προϋπολογισμό. Η Πέτρα είπε ότι δεν αυξάνει ο προϋπολογισμός όπως θα θέλαμε. Δεν γίνεται τριπλάσιος. Ο Όλαφ Σόλτς, ο Υπουργός ε, Οικονομικών, μέσα στη μεγαλοθυμία του, είπε ότι 1% αρκεί. Όχι, πρέπει να του πούμε του κυρίου Σόλτς, δεν αρκεί το 1% χωρίς μικρόφωνο. Η Πρόεδρος. Η Κομισιόν τώρα. Μια σύντομη αντίδραση. Συμφωνώ ότι το πρόγραμμα δεν αφορά μόνο τους φοιτητές. Πρέπει να αφορά και άλλους. Και προσπαθήσαμε να κάνουμε μια καλή πρόταση που να απεικονίζει αυτή την ιδέα ότι δεν καλύπτει μόνο τους φοιτητές το πρόγραμμα, ε, και αυτό ποιο είναι, ότι αν κοιτάξετε την έμφαση και το, την κατανομή του προπολογισμού θα δείτε ότι όλοι οι τομείς κερδίζουν, αλλά ειδικά ε, τα σχολεία, η νεολαία, η εκπαίδευση και η επαγγελματική κατάρτιση κερδίζουν περισσότερο. Ακριβώς για αυτό το σχόλιο που κάνετε και γιατί ακριβώς ε, κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης αυτά μας είπαν ενδιαφερόμενοι. Αυτοί οι τομείς έχουν ε, δυναμικό για να φτάσουν και την, να μας δώσουν και την κρίση μάζα, την οποία δεν έχουμε πετύχει σήμερα και αυτό είναι πολύ σημαντικό τμήμα. Σε ό,τι αφορά τις ε, πράξεις, κατεξουδότηση, εκτελεστικές κτλ. Ο ε, κανονισμός προτείνει κατεξουδότηση πράξη. για να ορίσουμε ειδικά τους επιπλέον δείκτες και το πλαίσιο παρακολούθησης. Αυτό προτείναμε εμεί, αλλά σε ό,τι αφορά την εφαρμογή πιστεύουμε ότι το τρέχον σύστημα ισχύει καλά, η εφαρμογή είναι ένα πράγμα. Εμείς έχουμε το πλαίσιο και την ε, εφαρμόζουμε και το εφαρμόζουμε με βάση το πλαίσιο. Είναι καλό αυτό το σύστημα, δεν θέλουμε να το προτείνουμε, να προτείνουμε κάποια αλλαγή του συστήματο αυτού. Εφαρμογή, δηλαδή πλαίσιο, συγγνώμη, και εφαρμογή. Μάλιστα, η Κομισιόν πιστεύει ότι κατεξουσιοδότηση και εκτελεστικέ πράξει και ειδικά οι εκτελεστικέ πράξει θα λειτουργήσουν καλά. Εντάξει, το καταλαβαίνω. Και εγώ, σαν πρόεδρο, θέλω να σα πω ότι θα με βόλευε πάρα πολύ να με ανακατεύεστε όλη την ώρα στη δουλειά μου αλλά δεν θα ήταν και τόσο ανοιχτή η συζήτηση. Ειδικά όταν τα πράγματα είναι λίγο αόριστα, οι εκτελεστικές πράξεις δεν είναι απλώς εκτελεστικές, είναι πολιτικές στην τελική φάση. Και βεβαίως εκεί θα πρέπει να εμπλακεί και το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. Άρα θα πρέπει να το ξανασυζητήσουμε το θέμα αυτό. Ο κύριος Φλίν. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Τρία σημεία. Πρώτον, Οποτεδήποτε συζητούμε το Εράσμος, ε, αισθάνομαι ότι υπάρχει και μια επιπλέον φιλοδοξία, την οποία δεν τη λέμε ξεκάθαρα, που είναι πέρα από την ε, προσπάθειά μας να υπάρξουν ανταλλαγές, φιλικές σχέσεις, πολιτιστικές ανταλλαγές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ότι προσπαθούμε να δημιουργήσουμε πολιτική υποστήριξη ε, στους πολίτες για την ε, ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Νομίζω ακούστηκε από τους πυρογνώμανες μας ότι το 83% των πολιτών που πηγαίνουν στα Εράσμους αισθάνονται περισσότερο Ευρωπαίοι. Εγώ θα ήθελα να πω ότι αυτό είναι επικίνδυνο γιατί είναι σαν να επιδιώκουμε την καταστροφή, την προοδευτική των, κρατών, των, κρατών, εθνών κρατών. Ε, μια, ε, κάτι προς το οποίο πολλοί αισθάνονται πολύ μεγαλύτερη και σημαντικότερη να ανήκουν πολύ περισσότερο. Κατά τα άλλα, άκουσα ότι θα προσπαθούμε να φτάσουμε και να απευθυνθούμε περισσότερο σε ανθρώπους ε, που να είναι πιο μειονεκτούντες. Ακριβώς επειδή το γεγονό ότι κανείς μπορεί να πάει σε μια άλλη χώρα και να σπουδάσει και να ζήσει εκεί, μπορεί αυτό να είναι ακόμα μεγαλύτερο, πιο σημαντικό και να αλλάξει τη ζωή κάποιου που μειονεκτεί. Και ότι με αυτόν τον τρόπο θα αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα στις κοινωνίες μας, οι οποίες δεν έχουν πια συνοχή, ακριβώς επειδή έχουμε ανθρώπους από άλλες κοινωνίες με διαφορετικές αξίες. Ελπίζω αυτό λοιπόν να το λάβουμε υπόψη μας. Τρίτον, αναφέρθηκαν διάφοροι συνάδελφοι στη θέση που θα έχει το Ηνωμένο Βασίλειο σε όλα αυτά. Και είπαν μάλιστα ε, και θα ήθελα μάλλον να επισημάνω ότι το Ηνωμένο Βασίλειο παράλληλα το γεγονό ότι φεύγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει μια μεγάλη δύναμη στον τομέα τη εκπαίδευση και τη έρευνα και πιστεύω ότι θα ήταν απαράδεκτο οι Βρυξέλλε να προσπαθήσουν να περιθωριοποιήσουν ή ακόμα και να αποκλείσουν το Ηνωμένο Βασίλειο από ένα τέτοιο πρόγραμμα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Δεν χρειάζεται να δώσω αμέσως... Α, απαντήστε θέλετε η τροπή. Να διευκρινίσω ότι οι συμμετέχοντες απαντούν ό,τι θέλουν. Και το 88% μας λέει ότι αυξήθηκαν οι γνώσεις τους, πάνω από το 80% μας λένε ότι έμαθαν ποιες είναι οι ευρωπαϊκές αξίες Επομένως αυτά είναι αυτά που οι ίδιοι συμμετέχονται στο Εράσμους μας απαντούν. Δεν είναι μια αξιολόγηση την οποία, στην οποία επισέρχεται η άποψη της Επιτροπής. Σας ευχαριστώ. Δύο λεπτά. Πιστεύω ότι το γεγονό ότι είχαμε 100% απορρόφηση του προπολογισμού δείχνει πόσο μεγάλη ήταν η ζήτηση. Γι' αυτό θα συμφωνήσω και με πολλού άλλου συναδέλφου ότι πρέπει να επιμείνουμε σε αυτό που έχει ζητήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τριπλασιασμό του προϋπολογισμού. Ακόμα περισσότερο, δεδομένου ότι τα χρήματα του Εράσμου θα καλύπτουν και άλλες δραστηριότητες συμπεριλαμβανομένες της πρωτοβουλίας ανακαλύπτοντας την Ευρώπη. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας όχι μόνο το ύψος των ποσών, αλλά ακόμα και το τι προβλέψεις, ε, ε, ε, επίσης τι προβλέψεις έχουμε για τον αριθμό των αιτήσεων. Πρέπει κανείς να δει υπό αυτό το πρίσμα το διπλασιασμό ή τον τριπλασιασμό του συνολικού προϋπολογισμού. Από τη μελέτη που μας παρουσιάστηκε, διαπιστώνω ότι υπήρξε υποστήριξη προς τον τομέα της νεολαίας και να ρωτιέμαι εάν θα υπάρξει μεγαλύτερη ε, υποστήριξη μάλλον στον τομέα του αθλητισμού. Αυτό το, γνωρίζω και από την επαφή μου με του νέου στη Μάλτα που θα ήθελαν περισσότερο να συμμετάσχουν στο Εράσμου, αλλά ιδιαίτερα από την πλευρά του αθλητισμού. Τώρα, όσον αφορά την ε, σχέση, την προσπάθεια που θα γίνει μάλλον να καταπολεμήσουμε τον αποκλεισμό και να φτάσει σε περισσότερους. Ε, ανθρώπους στο Εράσμος. Πιστεύω ότι πρέπει να κάνουμε δουλειά δημοσιότητας, έτσι ώστε να μην έχει αυτή την αίσθηση κανείς ότι το Εράσμος αφορά μόνο την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Εδώ τα πράγματα δεν θα είναι εύκολα. Όσον αφορά τώρα τη... τα άλλα προγράμματα, είπατε ότι θα μπορούν να αξιοποιηθούν χρήματα και από το Ευρωπαϊκό Επενδυτικό Ταμείο. Θα ήθελα να μου δώσετε περισσότερες πληροφορίες. Ε, γιατί θα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι το Εράσμος δεν θα απευθύνεται μόνο σε εκείνους που έχουν την οικονομική δυνατότητα, αλλά και, αλλά και σε εκείνους τους φοιτητές οι οποίοι δεν έχουν τα μέσα για να σπουδάσουν τα οικονομικά. Ένα άλλο ενδιαφέρον έβρεμα τη έρευνα είναι η ενίσχυση της πολυπολιτισμικότητας, αυτό το άνω του 80% των συμμετοχών που το αισθάνθηκαν Επομένως το ζήτημα δεν είναι μόνο να αισθάνεται κανεί περισσότερο Ευρωπαίος, αλλά να αυξηθεί επίσης και η ανοχή και η αντίληψη που έχει για τους άλλου πολιτισμού. Σας ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος, μιας και αναφέρθηκε δύο φορέ η έρευνά σας, κυρία Φαντεγκράφ. Σας ευχαριστώ για τις διαπιστώσει που κάνατε. Όσον αφορά τώρα το ζήτημα του αθλητισμού. Είναι ένας τομέας ο οποίος τώρα ξεκίνησε και θα πρέπει να δούμε την υλοποίηση του προγράμματος αργότερα. Όμως μπορώ να επιβεβαιώσω αυτό που είπατε ότι η ανταπόκριση των συμμετοχόντων ήταν θετική. Ήταν ε, περιορισμένη η παρέμβαση που είχε τη δυνατότητα να κάνει η Επιτροπή εδώ με τα χρήματα που είχε, αλλά κατάφερε πολλά, ιδιαίτερα στον τομέα των οργα... της βάσης των μικρών οργανώσεων λίγα στοιχεία έχουμε στη διάθεσή μας, αλλά τα λίγα στοιχεία που έχουμε επιβεβαιώνουν αυτό που λέτε. Και η αξιολόγηση ενδιάμεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο ίδιο συμπέρασμα καταλήγει. Στον αφορά τώρα στις ευάλωτες ομάδες. Συμφωνώ. Φαίνεται και στη νέα πρόταση της Επιτροπής το διαπιστώσαμε με χαρά ότι το Εράσμος δεν θα πρέπει να απευθύνεται σε εκείνους που θα τους ήταν εύκολο έτσι και αλλιώς να ταξιδέψουν, αλλά θα πρέπει να φροντίσει να είναι προσβάσιμο σε όλους. Και ε, τώρα, όσον αφορά τη συμπληρωματικότητα του Εράσμου με άλλα προγράμματα, όπως πιο συγκεκριμένα το πρόγραμμα επενδύσεων, αυτά θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να βελτιωθεί πρόσβαση. Για παράδειγμα, για τα ταξιδιωτικά έξοδα. Ε, ορισμένες, σε ορισμένε περιπτώσει υπολογίζονται ω ποσό κατά αποκοπήν, χωρί αυτό να ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Σε ορισμένε περιπτώσει το ταξίδι είναι πιο μακρινό. Ε, σε τέτοιες περιπτώσεις θα μπορούσε κανείς να χρησιμοποιήσει συμπληρωματικά άλλα ευρωπαϊκά κονδύλια, όπως για παράδειγμα αυτά που έχουμε τις επενδύσεις. Σας ευχαριστούμε για αυτές τις σημαντικές και ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις. Κύριε Έριξον, Επιτροπή. Σύντομα, μας ζητήσατε στοιχεία για τον αριθμό των συμμετεχόντων σε κάποια διάφορα προγράμματα. Μπορώ να σας δώσω κάποιες πληροφορίες. 12 εκατομμύρια είναι ο συνολικός αριθμός των δικαιούχων, 3 εκατομμύρια φοιτητές, 2 εκατομμύρια μαθητές 1,8 σπουδαστές στη μη τυπική εκπαίδευση και 3,6 6,3 εκατομμύρια ε, στην νεολαία. Ε, καθώς επίσης και 2 εκατομμύρια ε, δάσκαλοι και α, καθηγητές. Τώρα, όσον αφορά τον τομέα του αθλητισμού, θα διαπιστώσετε ότι πράγματι το, σε αυτό το τομέα έχει διπλασιαστεί ο προπολογισμό του διαθέσιμου κονδύλι. Επομένω, φαίνεται ότι ε, προσπαθούμε να συνεχίσουμε τις επιτυχίες που είχαμε στο πρόγραμμα Erasmus Plus. Θα διαπιστώσετε επίσης ότι προσπαθούμε να αυξήσουμε και την κινητικότητα των προπονητών και του προσωπικού του, που ασχολείται με τον αθλητισμό. Αυτό είναι επίσης ένα στοιχείο καταπολέμησης του αποκλεισμού, γιατί συχνά αυτές οι μικρές αθλητικές οργανώσεις έχουν στις τάξεις τους ε, παιδιά και νέους από μειονεκτούντες ομάδες. Τώρα, όσον αφορά την αξιοποίηση, τη συμμετοχή μάλλον τη μεγαλύτερη, και τη δημοσιότητα που θα χρειαστεί. Θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε με αθλητικές οργανώσεις, με οργανώσεις νέων, έτσι ώστε να μάθουν για το Εράσμους παιδιά που μπορεί να μην το είχαν σκεφτεί ως δυνατότητα. Ε, θα πρέπει να απευθυνθούμε λοιπόν σε αυτές τις κοινότητες, σε αυτές τις ομάδες, μέσω αυτών των οργανώσεων. Βέβαια, η καταπολέμηση του αποκλεισμού περνάει και από άλλα από άλλες προσπάθειες, θα πρέπει να γίνει μια επαναξιολόγηση του ύψους των επιδοτήσεων που δίνονται έτσι ώστε ε, να φροντίσουμε οι φοιτητέ και οι σπουδαστέ που δεν συνηθίζεται να συμμετέχουν στο Εράσμο αυτή τη στιγμή να το πράξουν. Ιδιαίτερα, για παράδειγμα, από μειονεκτούντε περιοχέ ή από μειονεκτούσε ομάδε. Τώρα, για τη σχέση με το ESF σε κάποιους τομείς νομίζω θα έχουμε μεγαλύτερη συνεργασία. Γνωρίζουμε ότι αυτή τη στιγμή είναι 70 εκατομμύρια οι ανεδικευτοί εργάτες στην Ευρώπη. Δεν θα μπορούσε το Εράσμος μόνο του να λύσει το πρόβλημα, αλλά εάν το δει κανείς ως συμπληρωματικό προς το ESF, μπορούμε να κάνουμε πράγματα. Μπορεί για παράδειγμα το ESF να χρηματοδοτήσει μετεκπαίδευση και το Εράσμος να έρθει να ασχοληθεί με το κομμάτι, για παράδειγμα, της διασυνοριακής συνεργασίας, της κινητικότητας των καθηγητών κτλ. Έτσι κάπως φανταζόμαστε τη σχέση των δύο προγραμμάτων. Σας ευχαριστώ. Και εμείς σας ευχαριστούμε, κυρία Κώστα. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η μελέτη και σας ευχαριστώ. Γιατί έχει και μια πολιτική και θεσμική διάσταση σημαντική για το Κοινοβούλιο. Ε, το ερώτημα που θέτεται στο τέλος. Δηλαδή ότι θα πρέπει να διευρυνθεί το πρόγραμμα σε επίπεδο με απόλυτων τιμών, ε, χωρίς αποκλεισμού και αυτό είναι κάτι που ενδιαφέρει το Κοινοβούλιο και θα το συζητήσει. Σε κάποια φάση λέτε ότι θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη διαβούλευση των τελικών αποδεκτών. Υπό ποια έννοια το λέτε αυτό, ποιοι είναι οι τελικοί αποδέκτες, γιατί η διαβούλευση ούτως ή άλλο. Σε ό,τι αφορά τα όσα είπε η κυρία Έριξον, το πρόγραμμα είναι πιο συνεπές με τη στρατηγική που ε, αναπτύξατε τα τελευταία χρόνια για την οικοδόμηση ενός ευρωπαϊκού χώρου εκπαίδευσης. Είναι ο βασικός στόχος. Τώρα, κάποιες διευκρινήσεις και μετά θα μιλήσω για τον προϋπολογισμό. Καταρχάς, για τη διαβίου μάθηση. Αυτή είναι μια μόνιμη αναφορά σε σχέση με τον νέο προϋπολογισμό και τους νέους πόρους θέλει να δώσετε μεγαλύτερη προτεραιότητα. Δηλαδή αλλάζουν τα ποσοστά ανάμεσα στα διάφορα προγράμματα. Ε, δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στους ενήλικες. Ε, βάζετε, βάζετε επίσης και, την, και τα μάστερ και τα ντοκτορά. Ε, επαγγελματική ε, κατάρτιση, νέους και στο τέλος βάλετε αυτό που σας ζητήσαμε. Ε, κινητικότητα των φοιτητών των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Σημαντικό αυτό. Επίσης, προσθέτεται και τα δίκτυα ευρωπαϊκών πανεπιστημίων. Όμως δεν υπάρχει πια ε, συγκεκριμένη αναφορά αυτή που υπήρχε στο Εράσμος Μούντος, που και όλα όσα προέβλεπε. Ξέρετε τώρα για τον προϋπολογισμό. Να επαναλάβω κάτι. Ναι, έχουμε αυξήσει κατά 26 δισεκατομμύρια. Ε, όμως θα αφαιρέσουμε τα κονδύλια του Discovery U, και αυτό είναι και το ερώτημά μου. Δεν υπάρχει πια αυτό που υπήρχε παλιά για τον εθελοντισμό. Έτσι, ε, φαντάζομαι κάπου αλλού πήγε, σωστό είναι αυτό. Τελευταίο, σε ό,τι αφορά κάποιες πρωτοβουλίες που είχαμε ζητήσαμε και που ε, επιβεβαίωσε ο κύριος Ναύρατσης, ε, η κάρτα για τους φοιτητέ. από πού χρηματοδοτείται. Τώρα, σε σχέση με τα άλλα προγράμματα, να μια στιγμή να τελειώσω, Πρόεδρε. Το θέμα των σχέσεων με τα διάφορα προγράμματα. Αυτό το λέμε για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Plus, για τον ορίζοντα. Υπάρχει σχέση με, αυτή, με αυτά τα προγράμματα. Με άλλα όμως δεν υπάρχει. Γιατί αν δεν υπάρχει σχέση με τα άλλα προγράμματα, λέει τι γίνεται. Κυρία Βάντεργκραφ, ε, θέλετε να απαντήσετε στις ερωτήσεις που σας αφορούσαν. Πρώτη, ναι, ότι θα πρέπει να προσεγγίσουμε περισσότερους δικαιούχους. Εγώ ως ερευνήτρια πάντα είμαι πέρα αυτού. Ε, πρέπει να μιλήσουμε με αυτούς τους τελικούς δικαιούχους σε οποιοδήποτε πρόγραμμα. Και πάντα σε οποιοδήποτε πρόγραμμα πρέπει να δοθούν να, γίνουν στοχεύσεις και να επιλέξουμε, να γίνουν επιλογές. Εγώ ε, μίλησα με κάποιου από του δικαιούχου, ειδικά σε κάποιε χώρε. ε, και πάντα είμαι υπέρ του περισσό, της ιδέας του περισσότεροι δικαιούχοι να υπάρχουν κτλ. Επίσης, ε, χάρη σε αυτές τις προσωπικές επαφέ, πήρα και κάποια στοιχεία, κάποιε αποχρώσεις που δεν θα τα είχα λάβει αν διάβαζα μόνο τη βιβλιογραφία. Για τα υπόλοιπα σχόλια δεν μπορώ να απαντήσω λεπτομερώς, δεν μπορώ να σχολιάσω. Είδαμε ότι οι εθελοντικές δραστηριότητες Α, δεν μπορώ να μιλήσω για αυτές. Θα μιλήσει η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το θέμα αυτό. Σας ευχαριστώ, κυρία Ρίξον, έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Ένα σημαντικό σημείο, πράγματι. Και να σας πω ότι οι διαβουλεύσεις πριν από την κατάθεση των προτάσεων, γιατί φυσικά λάβαμε ένα εκατομμύριο απαντήσει απαντήσεις και πολλές από αυτούς ήταν και από τους τελικούς δικαιούχους και πολλά από αυτά έχουν συμπεριληφθεί στις προτάσεις μας σήμερα, γιατί πραγματικά οι απαντήσεις μας έχουν να κάνουν με αυτά που μας είπαν οι δικαιούχοι. Σκεφτόμαστε λοιπόν ε, την προετοιμασία της εφαρμογής. Αυτό και κάνουμε τώρα. Και έχουμε καλή συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς και όλους όσους συμβάλλουν. Θα θέλαμε λοιπόν και αυτά να συμπεριληφθούν στην φάση προπαρασκευή. Θα πρέπει να βρούμε λοιπόν έναν τρόπο να διαβουλευτούμε και με τους τελικούς δικαιούχους και δεν έχω όμω σήμερα κάποιο συγκεκριμένο τρόπο να προτείνω. Συμφωνώ μαζί σας πάντως ότι είναι σημαντικό να υπάρχει τελικά πάντα κάπου στο μυαλό μας και ο τελικός δικαιούχος για τον εθελοντισμό. Όντως, ε, σωστή παρατηρήση που κάνετε. Όλες αυτές οι δραστηριότητε λοιπόν που περιλαμβάνονταν στην Ευρωπαϊκή Εθελοντική Διαδικασία μπορεί να περιληφθεί πλέον ε, στο Ευρωπαϊκό Σώμα άμα εθελοντισμού και αλληλεγγύηση αλλά να έχετε υπόψη σας ότι δεν έχουν χαθεί αυτά τα κονδύλια έχουν διπλασιαστεί και πλέον, δεν έχουν πάει χαμένα. Και επίσης ενδιαφέρουσε η παρουσίαση ότι το κόστος του αστραντισμού ήταν το πιο κοστοβόρο, άρα η αφαίρεσή τους βοηθά την υπολογισμό του τριπλασιασμού για να καταλάβετε που βρισκόμαστε. Ελπίζω να ήταν αυτό ε, ξεκάθαρο εξ αρχής, αλλά ουσιαστικά υπήρχε διπλασιασμό σε, σε όλα τα επίπεδα, σε όλους τους τομείς. Ε. Σε κάποιους τομείς χρειάστηκε κρίσιμη μάζα, και λίγο μεγαλύτερη αύξηση στον τομέα της ε, νεολαίας, της κατάρτισης, της εκπαίδευσης. Αλλά ναι, και η φοιτητική κάρτα Ε, κάνουμε μεγάλες προσπάθειες στην πλωτική αυτή φάση για να καταστεί λειτουργική από το 2021 αυτή η κάρτα από την έναρξη του νέου προγράμματος. Αυτός είναι ο στόχος μας. Μάλιστα. Ο κύριος Νέκοφ έχει το λόγο για δύο λεπτά. Ευχαριστώ, Πέτρα. Και θα ήθελα να καλωσορίσω την ομάδα από τη Βουλγαρία που περιλαμβάνει φοιτητέ από τον τομέα της ψηφιακής τεχνολογίας, κάποιοι από τα πορίσματα της μελέτης για την ε, μακροπρόθεσμη εκπαίδευση ως τα στοιχεία του Erasmus Άρα, στόχος είναι να περιληφθεί ένα 25% το πληθυσμό, 25 έως 65 και 25% να συμπεριληφθεί. Από αυτό το 25% ωστόσο, μόνο 4% του προγράμματος Εράσμους ε, από το Ερασμός ε, για τα άτομα 25 έως 65 χρονών καλύπτεται μόνο 11%. Στην Βουλγαρία το ποσοστό αυτό είναι κάτω από 2%. Πού πιστεύετε ότι ο προϋπολογισμός 4% του προγράμματος θα καλύψει 25% των ανθρώπων ηλικίας 25 έως 65 χρόνων με δραστηριότητες διαβίου μάθησης. Δεύτερη ερώτηση. κοινωνική φύσεω. Στην Ανατολική Ευρώπη έχουμε πολλά παιδιά από φτωχέ οικογένειε. Ακόμα και αν επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Erasmus Plus, πολύ απλά δεν μπορούν οικονομικά. Δεν θα βγάζουν πέρα. Σκέφτεστε μήπω ε, το ενδεχόμενο υψηλότερων υποτροφιών για τα παιδιά αυτά για να συμμετάσχουν στο Erasmus Plus. Ευχαριστώ, λέει η πρόεδρο. Κυρία Έριξον. Μάλιστα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ερώτηση και να καλωσορίσω και όλους τους ε, φοιτητέ από τη Βουλγαρία. Να συμφωνήσω λίγο γιατί μιλήσατε για τον εθνικό στόχο σε ό,τι αφορά την διαβίου Φυσικά πρόκειται για εθνική δέσμευση και το Erasmus Plus δεν μπορούμε να υποκριθούμε ότι θα βοηθήσει και θα λύσει το θέμα αυτό. Μπορεί να αποτελέσει ένα επιπλέον εργαλείο, αλλά αυτό προφανώς έχει να κάνει και με τις εθνικές προσπάθειες και τις εθνικές πολιτικές για την διαβίου μάθηση. Ελπίζω λοιπόν αυτό είναι σαφές, αλλά κοιτώντας το ποσοστό των νεαρών ανθρώπων Τώρα έχουμε χαμηλότερο ποσοστό από 4%. Ελπίζουμε με το νέο πρόγραμμα να είναι πάνω από 10% οι νέοι που ωφελούνται από το πρόγραμμα. Αλλά αυτά είναι εκτιμήσεις προφανώς. Δεν μπορούμε να τα θεωρήσουμε δεδομένα για τις μειονεκτικές ομάδες. Ναι, βεβαίως, είναι σημαντικό να κοιτάξουμε τα επίπεδα υποστήριξης, τα βασικά επίπεδα υποστήριξης. Να δούμε πώς μπορούμε να υποστηρίξουμε άτομα από μηνεκτικές περιοχές, αλλά δεν μπορούμε ασφαλώς να υποκαταστήσουμε και την εθνική αρμοδιότητα. Δεν πρόκειται... Δεν μπορεί να αντικαταστήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση την εθνική πολιτική και τις ανισότητες που υπάρχουν σε επίπεδο κρατών μελών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει πρόεδρος. Σε ό,τι αφορά την συμπερίληψη όλων, είναι σημαντικό. Γιατί ο τομέα της νεολαίας, σε ό,τι αφορά την άτυπη και ανεπίσημη εκπαίδευση και τις ε, διασυνοριακές ε, δραστηριότητες, για τους νέους που αντιμετωπίζουν μείον εκτήματα. Είναι σωστά αυτά που μας είπατε και έχω την εντύπωση ότι κυρίως σε ό,τι αφορά το θέμα της διαφοροποιημένης παροχής υποτροφιών η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάπως ε, νύπτει τα σχήρα της και λέει ότι τα κρατημέλη θα πρέπει να το καθορίσουν αυτό. Τώρα δεν ξέρω αν αυτό ήταν ο αρχικός μας στόχος για τη τελική ανάλυση. Θα παραμείνουν οι ανισότητες που υπάρχουν σε εθνικό επίπεδο. Αλλά να κάνω και μια ερώτηση προς τους εμπρεγνώμονες μας. Ε, τα τελευταία χρόνια διαρκώς ακούμε από τα κρατημέλη ότι ο τομέας ε, του πρώην προγράμματος Εκομένιος για τη συνεργασία μεταξύ σχολών και σχολείων. Ουσιαστικά στα πλαίσια στους κόλπους του Erasmus Plus ε, κάπως υποτιμήθηκε. Καταρχάς ε, δεν έλαβε την απαραίτητη σημασία και κατά δεύτερον ε, θεώρησαν πολλοί οι οποίοι προηγουμένως χρησιμοποιήσαν το πρόγραμμα κομμένιος ότι πλέον έχει καταργηθεί. Αυτό το διαπιστώσατε και εσείς ε, στην ε, έρευνά σας. Ότι στέρισε τελικά το πρόγραμμα Κομμένιου στους κόλπους του Erasmus Plus. Σε περίπτωση δε που ίσχυε κάτι τέτοιο, πώς σκοπεύουμε να το αλλάξουμε αυτό στο μελλοντικό πρόγραμμα, αν καταλήξουμε στα ίδια αποτελέσματα. Uh, thank you for that question. Um, well, I would have to... Σας ευχαριστώ. Η απάντησή μου σχετίζεται και με τα σχόλια που έκανε ο κύριος Νέκοφ. Πράγματι, αρχικά διαπιστώσαμε ότι σε κάποιες χώρες μας λένε ότι έγινε πιο δύσκολο να λάβει κανείς χρήματα για σχολεία γιατί έχουν δυσκολέψει οι αιτήσει, έχουν ε, αυξηθεί επίσης οι απαιτήσει, χρειάζεται να βρεθεί κανείς ένας ηγετικός εταίρος και να βρει και άλλους εταίρους. Ε, οι πιο μικρές ε, οργανώσεις ε, εκπαιδευτικές δυσκολεύονται και αυτό που συνήθως κάνουν είναι ότι προσλαμβάνουν ένα πρόσωπο το οποίο ασχολείται με αυτές τις αιτήσει. Για έναν πάρα πολύ απλό λόγο, όλες οι οργανώσεις που χρηματοδοτούνται από το Εράσμους πρέπει να υποβάλουν πάρα πολλά στοιχεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι λίγες λοιπόν οι λίγοι εκπαιδευτικοί οργανισμοί που έχουν τη δυνατότητα να κάνουν κάτι τέτοιο. Ε, από πλευράς διοικητικού φόρτου και ε, ακόμα περισσότερο δεδομένου ότι δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι η αίτησή τους θα στεφτεί με επιτυχία. Αυτό πλήττει περισσότερο οργανώσεις οι οποίες μπορεί να απευθύνονται στις πλέον μεκτούσες ομάδες, τα σχολεία λοιπόν αξιοποιούσαν πολύ περισσότερο το πρόγραμμα κομένιους. Φαίνεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προσπαθεί να ξαναδώσει έμφαση στην χρηματοδότηση των σχολείων με τη νέα πρόταση. Επομένως, η σύσταση δική μας από τη μελέτη είναι ότι χρειάζεται η διαδικασία των αιτήσεων να είναι πάρα πολύ πιο απλή και να μπορεί να απευθύνεται και σε οργανώσει, οργανισμούς διαφορετικών μεγεθών, ιδιαίτερα τι πιο μικρές. Σα ευχαριστώ. Ε, ευχαριστώ. Αυτό συνάδε και με αυτά που ακούμε διαρκώ από τους ε, εταίρους μας σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα, ότι σε πολλέ περιπτώσει τα πράγματα είναι υπερβολικά περίπλοκα, αλλά σε διάφορα τα σχολεία πιστεύω ότι και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να συμβάλλουν το λιθαράκι του προκειμένου οι δάσκαλοι, δασκάλες οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον τομέα των προγραμμάτων αυτών να το κάνουν όχι στον ελεύθερο χρόνο τους ανάλογα με την προσωπική τους ε, διαθεσιμότητα αλλά να έχουν ε, μια χρονικά προδιαγραμμένη περίοδο για την διεκπαιρέωση των εργασιών αυτών να μην είναι κάτι που κάνουν στον ελεύθερο χρόνο του διασκεδάση ή ένα ψυχή δάσκαλη. είναι δουλειά. Για αυτά που έχουν να διδάξουν και στους ε, νέους, σε ό,τι αφορά δηλαδή την ε, συνεργασία με τους δασκάλους. Δεν είναι κάτι το οποίο κάνουν εθελοντικά στον ελεύθερο χρόνο τους, είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να οργανώνονται χρονικά. Αυτά είναι τα όσα πρέπει να κάνουν και τα κρατημέλη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και έτσι σήμερα λοιπόν ολοκληρώσαμε τη συζήτηση αυτή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και την κυρία Φάντεγκράφα και την Έριξον που ήταν στην διαθεσία μας για ερωταπαντήσεις ε, για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. Νομίζω ότι ήταν καλή η ανταλλαγή απόψεων. Η Επιτροπή νομίζω ότι θα έχει υπόψη της πώς θα διαμορφωθεί η συζήτηση στο μέλλον. Θέλουμε να πούμε ναι στην ευελιξία, αλλά όχι με κάθε τίμημα. Και κυρίως όχι με το τίμημα να μείνει απ' έξω το Κοινοβούλιο σε ό,τι αφορά λήψη πολιτικών αποφάσεων. Δεν επιτρέπεται κάτι τέτοιο. Εμείς είμαστε αυτοί που πρέπει να θέσουμε πολιτικές προτεραιότητες. Δεν είναι δυνατόν ως κοινοβούλιο να δώσουμε λευκή επιταγή. Και απλά να διαθέσουμε τα κονδύλια και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αποφασίσει πώ θα επιτευχθούν οι στόχοι που έχουμε ορίσει με τα χρήματα που έχουμε στην διάθεσή μα. Δεν επιτρέπεται κάτι τέτοιο. Θα πρέπει να γίνει μια συζήτηση και αυτό το θέμα θα πρέπει να το συζητήσουμε. Υπάρχουν πολλά άλλα θέματα τα οποία θα συζητήσουμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με τους εμπειρογνώμονες και φυσικά όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς καλούνται να μας ε, πούν την απόψή τους για την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Τσφέρ, ω συζητητής, ε, θα ξεκινήσει τις εργασίες του και οι σκιώδεις ε, θα λεφτούν υπόψη και ελπίζουμε σχετικά γρήγορα να μπορέσουμε να συνεχίσουμε τις εργασίες μας στο θέμα αυτό. Ελπίζουμε μέχρι το τέλος της θητείας μας να έχουμε τα πρώτα αποτελέσματα. Ευχαριστούμε πολύ. Και έχουμε και άλλο ένα θέμα στην ημερήσια εντάξει. Ο κύριος ε, Λόκεγκάρτ είναι έξω. Τον χρειαζόμαστε όμως για το γενικό προϋπολογισμό γιατί είναι εισηγητής μας. Ευχαριστώ τους προσκεκλημένους μας. Και πιείτε και ένα καφεδάκι τώρα ή εν πάση περιπτώσει ό,τι επιθυμείτε. liebe Kolleginnen und Kollegen, ich würde gerne zügig weitermachen. Να συνεχίσουμε λοιπόν, συνάδελφοι. Μήπω τελειώσουμε και λίγο πιο γρήγορα. Φαντάζομαι ότι όλου σα ενδιαφέρει, γιατί, αύριο το, γιατί σήμερα το απόγευμα έχουμε και πάλι συνεδρίαση. Πάμε στο 11 λοιπόν τη ημερήσια διάταξη Γενικό Προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση για το Οικονομικό Έτο 2019. Ο εισηγητής μας ε, είναι ο Μόρτιν Λόκεγκαρτ και η προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών είναι 22 Ιουνίου στις 11 το πρωί. Και να σας υπενθυμίσω ότι είχαμε συμφωνήσει όλες οι τροπολογίες να καταταθούν στα αγγλικά. Ιδάλλως δεν προλαβαίνουμε να κάνουμε τις μεταφράσεις. Να δώσω το λόγο στον ε, Μόρτεν Λεκεγκάρτ να μας μιλήσει. Πέντε λεπτά. Okay, I'll try to manage. Thank you. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ όλους για την καλή συνεργασία και την πρόσφατη ε, γνωμοδότηση της ΚΑΛΤ ε, και τους τριμερείς διαλόγους όπου πήγαν όλα πολύ καλά. Ο, η εντολή για τον προϋπολογισμό θα μπει στη μερίσια διάταξη της Ολομέλειας του Ιουλίου. Τώρα που είδαμε την πρόταση για τον προϋπολογισμό του 19, πρέπει να κοιτάξουμε κυρίως τον προπολογισμό για τον ΓΙΑΜΑ, που μας αφορά για τον πολιτισμό. Φυσικά, ο τρίλογος ε, είναι σημαντικός για τις τροπολογίες και τώρα θα πρέπει να δούμε και τις συγκεκριμένες γραμμές του προπολογισμού. Θα ήθελα να κάνω λίγες ε, παρατηρήσεις για τον ίδιο τον προπολογισμό. Κάποια από τα βασικά θέματα είναι, καταρχά το Erasmus+, Plus, η αναθεώρηση του Πουδουπού πρότεινε 100 εκατομμύρια ε, επιπλέον για το Erasmus Plus για την περίοδο 2017-2020 ε, για να υπάρχει μεγαλύτερη ε, συμμετοχή. Και τα υπόλοιπα 26 εκατομμύρια θα πρέπει να δοθούν το 19. Η λογική της Κομισιόν ήταν να υποστηρίξουμε τα επιτυχημένα προγράμματα ενώ οι γραμμές για τον αθλητισμό χρηματοδοτούνται σωστά ε, το πρόβλημα είναι ε, τι γίνεται με την νεολαία, ε, με την επαγγελματική κατάρτιση. Τα 26 θα πρέπει να διαιρεθούν με βάση το 88% στην εκπαίδευση και την κατάρτιση, 23 εκατομμύρια και 12% νεολαία. Περίπου δηλαδή 3 εκατομμύρια. Σε ό,τι αφορά το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, θα ξέρετε ότι με τη συμφωνία του τριμερού διαλόγου τη περασμένη εβδομάδα, η Κομισιό ε, μετά από αυτήν έστειλε μια τροποποιημένη επιστολή και τροποποιημένο προπολογισμό για να λάβει υπόψη το τι συμφωνήθηκε στον Τρίλογο. Επομένω, υπάρχει αυτή η συμφωνία. Δεν υπάρχει λόγο να υποβάλουμε τροπολογίε. Σε ό,τι αφορά το Δημιουργική Ευρώπη και τα ΜΜΕ, επιπλέον 2 εκατομμύρια ε, πέρα από το πουδουπού έχουν δοθεί στα ΜΜΕ για να συνεχίσουμε την προπαρασκευαστική δράση της ΑΡΤΕ για τον υποτιτλισμό. Ε, Europe Facility. Όπως είπαμε στην κνομοδότηση, θα προσπαθήσουμε να επαναφέρουμε τα λεφτά που πήγαν στην πρωτοβουλία ε, για την Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια, να επιτρέψουν το 1,1 εκατομμύρια 18.04.101. Ε, Δράσεις ε, για τα πολυμέσα. 2,1 επιπλέον εκατομμύρια. Ε, γραμμή 09-05-05. Πέρα από τα λεφτά που είχε συμφωνήσει να δοθούν οι Κομισιόν, βασίζεται στις συζητήσεις που κάναμε με την, στην Επιτροπή για τα ευρωπαϊκά δίκτυα. Κάναμε πολλές συζητήσεις γι' αυτό και τώρα φαίνεται ότι κάτι πετυχαίνουμε. Στις συζητήσεις είδαμε ότι απλώς αυτή είναι η απαρχή. Θα πρέπει να έχουμε πιο ρεαλιστικούς προϋπολογισμούς. Εγώ θα έλεγα 4 με 5 εκατομμύρια. Ούτως ώστε να υπάρχει επιτυχία. Είναι μια αρχή όμως. Έχουμε κάτι στα χέρια μας για να δουλέψουμε. Να σας υπενθυμίσω επίσης ότι η πλήρης αναθεώρηση της, της πρικοδότησης που ζήτησε η Επιτροπή ΚΑΛΤ ε, θα πρέπει να απεικονιστεί και στον προϋπολογισμό. Αυτές είναι αρχικές παρατηρήσεις μου. Περιμένω τα σχόλιά σας και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η δικασία τον επόμενο μήνα. Μήνα. Σας ευχαριστούμε. Λουίτζι. Καταρχάς, ευχαριστώ τον ε, εισηγητή για την παρέμβασή του. Πιστεύω ότι σε γενικό βαθμό Μπορούμε να συμφωνήσουμε με τις θέσεις του. Θα προσπαθήσουμε να υποβάλουμε κάποιες τροπολογίες. Δεν μπορούμε να μην επιμείνουμε γιατί υπήρχε και στις κατευθυντήριες γραμμές του κανονισμού για τον προϋπολογισμό του 2019 και μια και μιλάει για κατευθυντήριες γραμμές ε, και επιβεβαιώθηκε από την ε, Επιτροπή για το Εράσμους. Δεν μπορούμε να υποχωρήσουμε σε σχέση με, την, ε, με το αίτημα για αντιπλασιασμό. επιμένουμε σε αυτό λοιπόν. Θα πρέπει να συνεχίσουμε να μιλάμε γι' αυτό. Όλοι λένε ότι είναι το καλύτερο πρόγραμμα. Έχει τη μεγαλύτερη προσθέμενη ευρωπαϊκή αξία. Επομένω και κάτι συγκεκριμένο. Α πούμε να κάνουμε και με τα οικονομικά δηλαδή. Δεύτερο θέμα. Για το θέμα τη δημιουργική Ευρώπη. Θα πρέπει να ξεπεράσουμε λιγάκι τα δύο εκατομμύρια που ανακτήσαμε. Γιατί ένα πρόγραμμα ε, χρόνια υποχρηματοδοτούμενο. Και την ίδια συζήτηση θα πρέπει να την κάνουμε και για την Ευρώπη, για τους πολίτες. Εδώ κάναμε μια εμβάθυνση στην Επιτροπή ε, και στην Ολομέλεια, συζητήσαμε το θέμα δηλαδή, όλοι συμφωνούμε ε, ότι το πρόγραμμα αυτό είναι πρόγραμμα κλειδί σε σχέση με τις προκλήσεις για το μέλλον, το μέλλον της Ευρώπης κτλ. Επομένως, μου φαίνεται ότι είναι και η ώρα να βάλουμε και τα απαραίτητα ποσά, ε, γιατί το πρόγραμμα έχει μεγάλες δυσκολίες. Το αποτέλεσμα τελικά ποιο είναι. Το είπαμε και χθε. Μιλάμε συνέχεια για τον πολιτισμό, αλλά τη στιγμή που φτάνει η στιγμή να υποστηρίξουμε τα προγράμματα πολιτισμού, δεν βάζουμε το χέρι στην τσέπη. Συμφωνούμε λοιπόν ως συνεισηγητή. α κάνουμε μια προσπάθεια, τη στιγμή που κάνουμε τις προτάσεις, να επιμείνουμε με πολύ αποφασιστικό τρόπο για τα οικονομικά. Ευχαριστώ, Έλγα. Πρώτα σου δώσω το λόγο να κάνω και σε σένα μια ερώτηση. Κατά πόσον έλεγξε, κατά πόσον ο ερθωτικός προπολογισμό που υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το, ταμείο, για το Σώμα αλληλεγγύη, ανταποκρίνεται αυτά στα οποία είχατε συμφωνήσει. Αν δεν το έχει ελέγξει, πε το μα και κάνε αυτόν τον έλεγχο, κάνε αυτό το τσεκ για να είμαστε σίγουροι. Έχει το λόγο. Ευχαριστώ, ευχαριστώ και τον Μόρτον. Να συμφωνήσω με όλα σχεδόν όσα ανέφερε. Να επικεντρωθώ σε δύο σημεία. Καταρχάς, ό,τι αφορά το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύη, δεν είχα χρόνο να το ελέγξω. Αλλά αυτό που ήθελα να σα πω πριν με ρωτήσετε είναι ότι θα το κοιτάξουμε και θα πρέπει να εξασφαλίσουμε στην Επιτροπή Προπολογισμού ότι έχουμε τα χρήματα. Αυτή ήταν η συμφωνία με την Επιτροπή. Και τώρα είναι καθήκον μας να ασκήσουμε πίεση για να συμβεί. Και θα σα πω, θα πραγματοποιηθεί. Αυτή ήταν η υπόσχεση της Επιτροπής. Να φροντίσουμε προκειμένου να πραγματοποιηθεί. Και νομίζω ότι 11 εκατομμύρια σε ένα χρόνο δεν θα πρέπει να αποτελέσουν πρόβλημα. Για το θέμα του ευρωπαϊκού του Ευρωπαϊκού Πολίτη και των επερχόμενων ε, εκλογών. Δίκιο έχει ο Μόρτεν. Θεωρώ ότι τα τις δραστηριότητες αυτές θα πρέπει να τις προωθήσουμε, όπως το Euronews για παράδειγμα. Είναι σαφές ότι χρειάζεται και το Euronews και το Euronet το Ευρωπαϊκό Ραδιοφωνικό Σταθμό. Θα πρέπει να αυξήσουμε, όχι να μειώσουμε τον προπολογισμό για να καλύπτουν όλο το ευρωπαϊκό Δικείο και είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί ενημερώνουν τον κόσμο στον σε κάθε κράτο μέλος, τι γίνεται σε άλλα κράτη-μέλη. Αυτό διαμορφώνει την πολιτική σφαίρα και γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να είμαστε σαφέστατοι προ το Συμβούλιο και την Επιτροπή ότι χρειαζόμαστε πιο πολλά χρήματα. Και ότι είναι προ το συμφέρον τους να αυξήσουν τον προπολογισμό και να υπάρχουν και καλέ δομέ στον Ωρανέτ και στο Euronews. Για το Ιρανέτ δεν νομίζω ότι αμφισβητήθηκε ποτέ. Για το Euronews έχει γίνει κάποια συζήτηση, αλλά αυτό που είναι σαφέ είναι το εξή. Αν δεν υπάρχει επαρκή ε, προπολογισμό, θα ψάξουν ιδιωτικό. Ιδιωτική χρηματοδότηση, γιατί δεν θα πρέπει να υπάρχει καμία παρέμβαση στο δικαίωμα διαμόρφωση του περιεχομένου. Είναι σαφέ λοιπόν ότι χρειαζόμαστε τα στοιχεία αυτά και στο Euronews λέει πρόεδρο διαπιστώνουμε ότι έχουμε και το κόστος τη μετάφραση. Μετάφραση σε πολλέ χώρε όπου θεωρούμε ότι είναι απαραίτητο να υπάρχει εκπομπή των προγραμμάτων αυτών. Αλλά τα προγράμματα αυτά δεν ε, μεταφράζονται, για παράδειγμα, στην Ικρανία. Μήπως να κοιτάξουμε ιδιαίτερα στην περίπτωση της Euronews αυτά που θέλουμε να πετύχουμε με τους πόρους τα πετυχαίνουμε. Δεδομένων και των ιδιωτικών ε, ιδιοκτησιακών δομών, το οποίο δεν είναι φυσικά καθε αυτό απορριπταίο, αλλά φυσικά υπάρχει η προσδοκία του κέρδους. Λογικό είναι. Να δούμε λοιπόν κατά πόσον αυτά που θέλουμε να πετύχουμε με τη χρηματοδότηση τα πετυχαίνουμε. Αμφιβάλλω. Κυρίως ό,τι αφορά και την ανεξαρτησία. Την ανεξαρτησία στον τομέα της σύνταξης στην Euronews. και τα προγράμματα όπως το Euronet Plus, όπου μιλάμε για προώθηση προγραμμάτων ή τα προγράμματα της ΑΡΤΕ με τις απαραίτητες μεταφράσεις. Φτάνει και αγγίζει μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού, 80% νομίζω. Μήπως έχει καλύτερα αποτελέσματα. Δεν ζητάει κανείς το λόγο. Θα δώσω λοιπόν το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας πει αν έχει οποιαδήποτε σχόλιο παρατηρήσει να κάνει. Όχι, από ό,τι φαίνεται. Μόρτεν. Well, thank you very much. And just, uh, Σας ευχαριστώ. Να ευχαριστήσω και τους Σκιώδης. Περιμένω τις τροπολογίες τους. Να κάνω κάποιες μικρές παρατηρήσεις για αυτά που ακούστηκαν. Σε μεγάλο βαθμό συμφωνώ και τα υποστηρίζω. Και το πρόγραμμα για τη Δημιουργική Ευρώπη και το Connecting Europe είναι σημαντικά στοιχεία του προπολογισμού. Το ίδιο συζητούμε εδώ και πολλά χρόνια. Και πιστεύω ότι είναι σημαντικό ως ε, Επιτροπή ε, από κοινού να συνεχίσουμε να επισημαίνουμε τη σημασία αυτών των προγραμμάτων. για να πιέσουμε το Συμβούλιο και την Επιτροπή να κάνουν τη δουλειά που πρέπει, δηλαδή να βρουν τα χρήματα που χρειάζονται. Θα πρέπει λοιπόν να επιμείνουμε σε αυτές τις αλλαγές στον προϋπολογισμό που προτείνουμε. Υποστηρίζω λοιπόν πλήρως αυτό που είπε ο Ιαν. Όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Σώμα Λεγγύης, θα παρακολουθήσουμε στενά τις εξελίξεις. Συμφωνώ πλήρως με αυτά που ακούστηκαν και είμαι σίγουρος και εσείς Χάνα θα κάνετε ό,τι πρέπει για να ε, διασφαλίσετε τα απαιτούμενα χρήματα. Ας έχουμε λοιπόν και εμείς το νου μας. Πολύ σημαντικό είναι αυτό που είπατε στο τέλος και εσείς κυρία Πρόεδρε. Πρέπει να δούμε τη δομή αυτών των προϋπολογισμών. Έχω συζητήσει με τους επακεφαλείς αυτών των υπηρεσιών και με τώρα πώς λειτουργεί η χρηματοδότηση. Χρειάζεται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως Κοινοβούλιο να έχει μια πιο αν θέλετε, χρηστή μέθοδο στην χρηματοδότηση αυτών των ε, δραστηριοτήτων. Είναι ε, συζητήσεις που είχαμε ξεκινήσει και παλιότερα και χρειάζεται να τις συνεχίσουμε. Το ίδιο ισχύει και για το Euronet Plus και για την πρωτοβουλία του Άρτε. Εδώ είναι πρωτοβουλίες τις οποίες θα πρέπει να προηγηθεί μια πολιτική συζήτηση για τις προτεραιότητες που έχουμε τη στιγμή που πλέον θα γνωρίζουμε ποια χρήματα, πόσα χρήματα είναι διαθέσιμα συνολικά. Ε, ελπίζω ότι συνολικά θα μπορέσουμε να αυξήσουμε το διαθέσιμο, τον διαθέσιμο προπολογισμό για όλες αυτές τις ε, πρωτοβουλίες, γιατί όπως είπατε τις χρειαζόμαστε. Ακόμα περισσότερο δεδομένου ότι έρχονται και οι ευρωεκλογέ. Και είναι στιγμή να το πούμε αυτό δυνατά. Αυτά από την πλευρά μου κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Ja, vielen, vielen herzlichen Ευχαριστώ. Και έτσι ολοκληρώσαμε την ε, πρώην μα συνεδρίαση για σήμερα. Μα εκεί γιατί λέει η πρόεδρο, ε, ότι θα ολοκληρώναμε μέχρι τι 12.30. Νομίζω ότι όλοι είμαστε ικανοποιημένοι. Έχουμε λίγο παραπάνω χρόνο το μεσημέρι. Και να σα υπενθυμίσω ότι στι 22 Ιουνίου στι 10 το πρωί έχουμε την προθεσμία που άλλαξε για τον προϋπολογισμό στα αγγλικά. Σας ευχαριστούμε Μόρτον και καλή συνέχεια στις εργασίες σας. Τα λέμε πάλι σήμερα το απόγευμα στις 3 για να συζητήσουμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη. Ελπίζω να τα πούμε το απόγευμα. Λοιπόν, καλό μεσημεριανό. Τα λέμε αργότερα.